Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εξωτερικών. Περνώ στο πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης, έγκριση. Εάν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνετε. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Και έτσι περνάμε στο σημείο 3 δημόσια κρόαση, προοπτικές της Λιβύης στην ε, περιφερειακή τρέχουσα κατάσταση. Καλώς ορίζω τους προσκεκλημένους μας και εκ μέρους του κυρίου Παντσέρη, πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα συμπροεδρεύσει. Καλώς ορίζω τους προσκεκλημένους λοιπόν τον κύριο Μοχαμέτ Φαχάτ, αναπληρωτή διευθυντή της αντιπροσωπείας της Λιβύης, αλλά και τον κύριο Μέστρα του Κέντρου του Ατλαντικού Συμβουλίου, ο κύριος Ματία Τουάλντο, ο οποίος ε, έχει προβλεφθεί για την, ε, για την ε, δημόσια αυτή ακρόαση, δεν θα μπορέσει να προσέλθει. Είναι γνωστή η κατάσταση στη Λιμβύη, την έχουμε συστήσει πολλές φορές. Είναι εύθραστη πολιτικά και σε επίπεδο ασφάλειας η κατάσταση. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης που υπογράφηκε πριν από δύο χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί λόγω των εσωτερικών αντιπαραθέσεων στη Λιβύη και δεν είναι γνωστό αν θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία οι πλευρές. Υποστηρίζουμε τη διαδικασία συμφιλίωσης στη Λιβύη των Εθνών που υποστηρίζουν ε, και την πολιτική συμφωνία και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις των προσκεκλημένων μας για τις προοπτικές του σχέδιου των Εθνών και την πορεία περαιτέρω. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που θα οδηγήσει σε νέα δεινά τους πολίτες και θα θέσει κίνδυνο τις ε, δυνατότητες για μια ε, πολιτική συμφωνία στην περιοχή. Η σταθεροποίηση της Λιβύης και η περάτωση της σύγκρουσης είναι κέρια σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και τη Μεσόγειο. Εν προκειμένου η περιφερειακή διάσταση έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς πολλοί είναι οι παράγοντες που έχουν συμφέροντα αλλά και διακυβεύματα στην περιοχή, ε, πολλά γειτονικά κράτη, αλλά βεβαίως όλο και περισσότερο εμφανίζεται ο ρόλος της Ρωσίας. Πριν ε, δώσω το λόγο λοιπόν στους ομιλητές, και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρο Ταγιάννη έχει ανακοινώσει επίσκεψη των Ευρωβουλευτών στη Λιβύη μέχρι το τέλο του έτου. Θα συντάξει μάλιστα σύσταση η ΑΦΕΤΑ για την Λιβύη με εισηγητή του συνάδελφο κύριο Παντσέρη. Και τώρα δίνω το λόγο στους προσκεκλημένους μας με τον αναπληρωτή διευθυντή τη ε, αντιπροσωπεία τη Λιβύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριο Μοχάμετ Φαρχάτ, και μετά θα πάρει το λόγο ο κύριο Καρή Μεσράν. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά μεγάλο τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε την ε, σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Λιβύη αυτή τη στιγμή. Όσοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγες τη εξελίξη ε, στη Λιβύη από το 2011, βλέπουν τα χαρακτηριστικά μιας ε, χώρας που βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε διάδοση των όπλων, των ενόπλων ε, δυνάμεων, κατακραματισμός ε, των κρατικών θεσμών, διαφθορά, οικονομική κρίση και η διαδοχή κυβερνήσεων δεν έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν την δημοκρατική μετάβαση λόγω της ε, πολιτικής πόλωσης που δημιουργήθηκε με τη μορφή των αμοιβαίων αποκλειούμενων ε, ομάδων. Εξαιτία των εσφαλμένων αποφάσεων, που ήταν πολλέ από τι προηγούμενε κυβερνήσει που συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού των ενόπλων ε, ομάδων που κατασπαταλούν το, τα, τα δημόσια κονδύλια. Το 2014 περάσαμε στην ένοπλη σύραξη και στην ανατολική και στη δυτική πλευρά της χώρας μας, που ε, ουσιαστικά χώρισε στη μέση τους ε, θεσμούς. και κάθε πλευρά ε, βασιζόταν σε διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις ε, η μία πλευρά τον, στον οδικό χάρτη του Φεβρουαρίου. Το κάθε νομοθετικό όργανο δημιούργησε τη δική του κυβέρνηση και οι δύο κυβερνήσεις ε, προσπαθούσαν να δυσφαλίσουν τον έλεγχο ε, ιδίως σε φορά τον Διεθνή Οργανισμό του Πετρελαίου και άλλους φορείς και δημιουργήσουν έτσι δύο φορείς για κάθε τομέα. Όπως ξέρετε, τα Ηνωμένα Έθνη μέσω των ειδικών αναπεσταλμένων έχουν προσπαθήσει ε, να καταλήξουν σε συμφωνία και να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των ε, λιβικών ε, θεσμών για να διαμορφωθεί η νέα κυβέρνηση. Ο κ. Μετσαλέμι είναι ο τρίτος που το ανέλαβε αυτό μετά την υπογραφή της Συμφωνίας 2015. Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του το περασμένο Σεπτέμβριο να τροποποιήσει την Λιβική Πολιτική Συμφωνία ζήτησε μια εθνική συνδιάσκεψη ε, και μετά εκλογές. Έχει υποβάλει λοιπόν πρόταση για αυτό που αποκαλεί μια πρόταση εκτελεστική εξουσία. Μετά από δύο έντονου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο ε, επιτροπών διαλόγου που εκπροσωπούν το HOR και ε, το Συμβούλιο τη Επικρατεία έγινε μία συνεδρίαση των, ε, όπου υιοθετήθηκε αυτή η πρόταση, ενώ το ε, Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα την έγκρισή του. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα και ανοριμότητα που πάντα αποτέλεσε εμπόδιο για τους διαμεσολαβητές προκειμένου να συνάψουν μία πολιτική συμφωνία. Επίσης, οι μηχανισμοί διαμεσολάβησης δεν έχουν εργαλεία άσκησης πίεσης και έτσι περιορίζονται σε ό,τι αφορά την άσκηση επιρροής. Για ό,τι αφορά την νομοποίηση των ε, οργάνων που προκύπτουν από την ε, συμφωνία αυτή, ε, κάποιοι θεωρούν ότι μία περίοδος Ε, δύο ετών πρέπει να παρελθεί ε, μετά από τον φετινό Δεκέμβριο. Υπάρχουν πιο περίπλοκα σενάρια όπου κάποιες πολιτικές ακόμα και ένοπλες δυνάμεις ε, θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να κερδίσουν έδαφος. Μπορεί να υπάρξουν νέες πολιτικές συμμαχίες, άλλοι φορείς μπορούν να αναλάβουν δράση, αλλά όχι με μια ξεκάθαρη δέσμευση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του σχεδίου. Ταυτόχρονα όμως η Λιβύη πρέπει να ε, επιτύχει πολιτική λύση και να ε, ενωθούν και πάλι οι κατακαιρματισμένοι θεσμοί της. Αυτό θα επιτρέψει πρώτα απ' όλα την επανένωση των ενόπλων δυνάμεων, ιδίως των τακτικών και οργανωμένων ή αυτών που ε, θέλουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης των κρατικών θεσμών. Και για να έχουμε αποτελέσματα πρέπει πραγματικά να υπάρξει ε, ανάκτηση του ελέγχου των ε, όλων των συνόρων, ε, προστασία των υποδομών και σημασία, των ευραλικών υποδομών και των ενεργειακών υποδομών. Θα θυμάστε πως έχουν κλείσει ορισμένα ορισμένες σταθμοί άντλησης πετρελαίου εδώ και χρόνια και κάποιες ομάδες ακόμα προσπαθούν να εκβιάσουν ε, το κράτος για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Μια μικρή ένοπλη ομάδα πρόσφατα έκλεισε υποδομές ε, παροχής νερού σε μικρές πόλεις δύο φορές με 45 μέρες για να ασκήσουν πίεση για την απελευθέρωση ενός ε, κρατουμένου στην Τρίπολη. Δεύτερον, θα επιτρέψει την εφαρμογή δέσμης μεταρρυθμίσεων για, κυρίως για τον έλεγχο των ε, δημοσίων δαπανών. Η σημερινή οικονομική κρίση έχει ασκήσει πίεση στους ε, πολίτες, ε, συνεχίζει να υποτιμά το νόμισμα με μεγάλο πληθωρισμό. Οι πολίτες μένουν στα ATM για ώρες για να πάρουν ρευστό η ανεργία έχει περιβεί το 20% και έχουμε πολλές οικονομικές παρατυπίες. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη ε, για νέο σχέδιο προπολογισμού με νέες μεταρρυθμίσεις και αυτά είναι πολύ σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη το σωρευτικό έλλειμμα το οποίο υπερβαίνει το 200% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος που έχει φτάσει τα 700 δις ε, λιβικά δινάρια φέτος, πέραν των όσων δαπάνησα η κυβέρνηση του HOR, που επίσης ε, υπολογίζεται στα 20 δισεκατομμύρια δινάρια. Τα αποθεματικά έχουν πέσει στα 47 ε, δις δινάρια και τρίτον η συνέχιση αυτής της, ε, η επανένωση μάλλον ε, της κυβέρνησης θα ε, μας βοηθήσει να στηρίξουμε τα έργα του Εθνικού Συμβουλίου Πετρελαίου για να επανέλθουμε στην παραγωγή ικανότητα του 1,6 εκατομμυρίου βαρέλια την ημέρα. Κυρίω τώρα σε ό,τι αφορά τι υποδομέ και τη στέγαση, ε, την ανοικοδόμηση πόλεων όπως το βγάζει. Πέμπτον, υλοποίηση προγραμμάτων DDR-SSR σε εθνική κλίμακα, καθώς αυτά τα προγράμματα δεν έχουν προωθηθεί στη Λιβύη από το 2011 και ε, απαιτούνται προγράμματα απενεργοποίησης ναρκών ε, σε σχεμένες πόλεις. Μετά συνέχιση της ε, πάλης κατά τρομοκρατικών δυνάμεων που παραμένουν και θυλάκων συγκεκριμένα. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν, θα επιτρέψουν την κυβέρνηση ε, να αντιμετωπίσουν τέτοια κέρια ζητήματα όπως είναι η εθνική συμφιλίωση, η επιστροφή των ε, εκτοπιστέντων ε, στα σπίτια τους, η στήριξη των δήμων και κοινοτήτων σε όλο αυτό το νέο εγχείρημα, καταπολέμηση της εγκληματικότητας που οφείλεται στην έλλειψη των αρχών επιβολής του νόμου σε κάποιες περιοχές είχαμε απαγωγές ε, για λίτρα και άλλες εγκληματικές δραστηριότητε και πάλι εξαιτία της ε, κακής ε, λειτουργίας του ποινικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ας περάσω τώρα στη μετανάστευση στη Λιβύη. Υπό το φως των τελευταίων εξελίσεων στη μεταναστευτική πραγματικότητα η Λιβύη στην ουσία αντιμετωπίζει το φαινόμενο πολλών βορειοαφρικανών να συγκεντρώνονται στις περιοχές γύρω από τα αστικά κέντρα στην, της Τρίπολης και η έκθεση αυτή η ενδιάμεση είναι κάτι βέβαια το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί και βάση περιπτώσει τα ευρήματα οφείλονται και στην οικονομική αδυναμία του κράτους να αντεπεξέλθει όπως επίσης και στις δραστηριότητες αυτών που εμπορεύονται ε, το ε, ανθρώπινο αυτό δυναμικό όπως και λόγω της αδυναμίας που έχει η Λιβύη να ελέγξει τα νότια σύνορά της δεν είναι σε θέση να ανακόψει την ροή των μεταναστευτικών ρευμάτων, ρευμάτων από τις ε, υποσαχαρικές περιοχές ο αριθμός των, των πληθυσμών υπομετακίνηση και εκτοπισμένων πληθυσμών έχει ξεπεράσει την Μέση Ανατολή. Άνω των 4 εκατομμυρίων κατοίκων των χωρών αυτών έχουν προσφύγει στις βορειότερες χώρες κοντά στη Μεσόγειο. Ε, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, ο πληθυσμός, τα δημογραφικά στοιχεία έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης στον κόσμο και η αγορά εργασίας στην Αφρική τα επόμενα 20 χρόνια θα χρειάζεται τη δημιουργία 20 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ετήσια για να αντιμετωπίσει τη ζήτηση. Η Λιβύη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μετακινήσεις αυτές και παρά τα δύσκολα επτά χρόνια που προηγήθηκαν η Λιβύη σε καμία περίπτωση δεν θέλησε είτε να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις ή να φτιάξει αναχώματα ελεγχόμενα στα νότια σύνορα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Λιβύη είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους όσο περισσότερο γίνεται έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των μεταναστευτικών κρίσεων και μέσω των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρώπης και στα πλαίσια των μέτρων έρευνας και διάσωσης τα οποία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μεσόγειο. Η στάση αυτή είναι λίγο θα έλεγα επιπόλαια και δεν παρέχει προστασία πραγματική στους μετανάστες οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς ούτε στην ίδια τη Λιβύη. Η διαχείριση λοιπόν των μεταναστών στην Λιβύη θα πρέπει να είναι τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου. Η χώρα μου έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει και όχι μόνο τη μετανάστευση. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ιταλία τώρα και η Ελλάδα έδειξαν ότι μπορούν να τύχουν υψηλού επίπεδου αλληλεγγύης από τις ευρωπαϊκές αρχές. Το ίδιο και οι αρχές στη Λιβύη. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε οι υπαρξιακές προκλήσεις, αλλά δυστυχώς η Αφρικανική Ένωση δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου. γίνονται ε, εκθέσεις από την συγκεκριμένη οργάνωση που χαρακτηρίζουν την χώρα μου κέντρο εγκληματικών δραστηριοτήτων και δουλείας, ενώ βέβαια η δουλεία ξέρουμε ότι υπάρχει κυρίως κατά τη διάρκεια της, ε, της οδού προς τη Λιβύη, κυρίως όμως από τις χώρες καταγωγής. Συνεπώς λοιπόν τα πράγματα εξαρτώνται από το πότε θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το κράτος στη χώρα αυτή, από πότε θα αποκαταστήσουμε την τάξη και το κράτος δικαίου στις περιοχές, στα σύνορα με την υποσαχαρική Αφρική. Είναι μια χώρα η Λιβύη με τεράστιους φυσικούς πόρους, μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις ε, απασχόλησης και για Λιβύους και για τους υπόλοιπους Αφρικανούς και νομίζω ότι η βοήθεια για την ανάπτυξη θα βοηθήσει τη χώρα μου, θα βοηθήσει και την ε, ε, υπόλοιπη περιοχή. Ένα προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς θα ευνοήσει την αλληλεία, τη γεωργία, την παραγωγή των τροφίμων και την προώθηση ε, εξαγωγών προς την Ευρώπη και αυτό θα βοηθήσει πολλούς νέους να βρουν εργασία στις λιβικές αγορές. Ε, δεν ξέρω αν οι, ε, τα μέλη της Επιτροπής σας θέλουν να θέσουν ορισμένες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακούμε τον κύριο Μεζράν. Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Ευχαριστώ τον κύριο Φαρχάτ για τα λόγια του. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα όσα μας είπε. Είναι σημαντικό να γίνουν αντιληπτά κάποια σημεία. Η κατάρρευση μετά την επανάσταση του 2011 της Λιβύης έχει πολλά αίτια, τα ερευνούν οι ειδικοί. Πολλά ανάγονται στην ιστορία της χώρας, που έτσι σε διαιρεμένη δεν ενώθηκε ποτέ, διαφορετικές ταυτότητες και πολλά άλλα. Άλλα έχουν να κάνουν με το καθεστώς του Καντάφη, πιο πρόσφατα αίτια, τον τρόπο της διακυβέρνησής του, το σύστημα του διέρη και βασίλευε, με την ιδέα της αποδυνάμωσης ταυτότητας των Λιβύων μέσα από την επιβολή της ιδέας του παναραβισμού. Αλλά υπάρχουν και πιο πρόσφατα αίτια. Τα δύο προπατορικά αμαρτήματα της Επανάστασης θα τα ονομάσω. Πρώτον, το ότι δεν έγινε αντιληπτό πως δεν επρόκειτο για επανάσταση λαού εναντίον δικτάτορα και μερικών μισθοφόρων, γιατί είχε σχηματίσει συνένεση γύρω του ο Καντάφη, είχε κόσμο που τον υποστήριζε από τον ε, πληθυσμό και το ότι αυτό δεν αναγνωρίστηκε και ότι καταδικάστηκε αυτό το γεγονός ε, οδήγησε στο ότι η λιβυική ελίτ υποτίμησε την σημασία των γεγονότων, ε, έσπευσε να κάνει εκλογές χωρίς να αντιληφθεί ότι χρειάζεται η επανασυμφιλίωση πρώτα να λάβει χώρα, ε, η επανένωση, ο προσδιορισμός του τι θέλουν οι πολίτες για τη Λιβύη. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα όσα θα σας αναφέρω αργότερα. Το δεύτερο προπατορικό αμάρτημα ήταν ότι η ξένη επέμβαση περιγράφηκε ως μια ελαχίστων διαστάσεων. Ε, Έγινε προβολή ιδιαίτερα του ρόλου των πολιτών, του απλού του λαού που κατέβηκε στους δρόμους και υποβιβάστηκε ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Και αυτό οδήγησε σε μια άμεση απόρριψη του ρόλου του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο μετά την Επανάσταση. Και αυτό πλέον όλοι το παραδέχονται. Σε περίπτωση βέβαια νίκη θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τον ΝΑΤΟ να παραμείνει στη Λιβύη, να αφοπλίσει τις ε, πολιτοφυλακές, να βοηθήσει στην επανασυμφιλίωση, εν πάση περιπτώσει να βγει ομαλά από τη χώρα, αλλά δεν συνέβη αυτό. Αυτά τα δύο προπατορικά αμαρτήματα οδηγούν σε μια καταδίκη της χώρας εξ αρχής, σε, μια, ένα κικαιώνα αταξίας, μαζί με τα... Ε, σφάλματα των κυβερνήσεων όπως αυτής του ΚΥΠ η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη των πολιτοφυλακών, την ε, διάδοση της δράσης τους και έριξε έτσι τους σπόρους μιας διαρκούς ε, ιστορικής σύγκρουσης. Το 2014 εκδηλώθηκε η έκρηξη με την ε, επιχείρηση του στρατηγού Χαφτάρ την επιχείρηση Καράμ ε, στην Μπενγάζη που απείλησε την Τρίπολη, ξέρετε πολύ καλά τι ακολούθησε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να πέσουμε στην ε, παγίδα ενός αφηγήματος που φέρνει ε, αντιμέτωπους τους υποστηρικτές ενός κοσμικού λαϊκού κράτους έναντι των Ισλαμιστών. Δεν είναι αυτό το πραγματικό αφηγήμα. Τα πραγματικά αίτια του, του διχασμού είναι ότι υπάρχουν οι Λίβοι που θεωρούν ότι ίσως δεν θα ήταν και τόσο άσχημο να επανέλθουν στο παλαιό καθεστώς μείον τον Καντάφη, στην παλιά μορφή διακυβέρνησης που είχαν, και εκείνων των δυνάμεων που είχαν πιο επαναστατικές βλέψεις και έλεγαν όχι, εμείς θα προχωρήσουμε προς το διαφορετικό. Και οι δύο πλευρές εκφράζονται και στα δύο μέτωπα της σύγκρουσης, και αυτό είναι εύκολο για να καταλάβουμε την κατάσταση, είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε την κατάσταση, αλλά υπάρχουν και στη μία πλευρά και στις δυνάμεις του Χαφτάρ αλλά και στην άλλη πλευρά, στου Σαράζ κτλ. Και αντίστοιχα υποστηρικτές του κοσμικού κράτους και στη μία και στην άλλη πλευρά. Οι φιλελεύθεροι αν θέλετε να τους πείτε έτσι. Και στα δύο μέτωπα και στα δύο στρατόπεδα. Αυτό για να καταστεί σαφέ ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μία μονολυθική και ομοιογενή ομάδα που, είναι, ε, που αντιπαλεύεται μια άλλη μονολυθική και ε, ενιαία ομάδα. Ωστόσο τα δεινά του λιβικού λαού έχουν φτάσει σε αφόρητα επίπεδα, υπάρχουν πολλοί φόβοι δεδομένοι και διάχυτη σε όλο τον κόσμο, το επίπεδο ζωής, ε, διακοπές ρεύματος, ε, ε, πληθωρισμός, απουσία ρευστού στην οικονομία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει κανείς να ζει υπό μαλές συνθήκες στη Λιβύη αυτή τη στιγμή και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο ε, αν θέλει κανείς να διαφυλάξει τη μετάβαση της Λιβύης, αν θέλει να διαφυλάξει το όραμα μιας χώρας με, ένα πλουραλιστικό σύστημα, που δεν θα το ονομάσω καν δημοκρατία, αλλά ένα ανοιχτό σύστημα, εν πάση είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα να δράσει ενωμένη πίσω από το σχέδιο των ΗΠΑ Εθνών, ταχύτατα και ενωμένη. Και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, γιατί χάνουμε το λαό της Λιβύης γίνεται πλέον, πέφτει σε μια απάθεια ο λαός, ε, παίρνει αποστάσεις, λέει καλά δεν πειράζει και ο Καντάφη να γυρίσει πίσω και αυτόν θα τον δεχθούμε. Εκεί έχει φτάσει και εδώ έχουμε την αρχή του τέλους, αν δεν δράσουμε γρήγορα, αν δεν μπορούμε να ξανακερδίσουμε τους πολίτες για το πολιτικό χώρο, να τους ε, καταστήσουμε πρωταγωνιστές, να τους δώσουμε ελπίδα, να τους πείσουμε να αγωνιστούν, να συμμετάσχουν, να εργαστούν σκληρά όπως είχε συμβεί στον πρώτο καιρό μετά την Επανάσταση, θα έχουμε χάσει αυτό το στοίχημα. Βεβαίως από το 2014 ξεκίνησε η διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και δεν πρόκειται εγώ να σας πω ότι στην θεωρία της διαπραγμάτευσης όταν υπάρχει στασιμότητα μεταξύ των δύο πλευρών που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στην ίδια κατάσταση, τότε έρχεται η ώρα της διαμεσολάβησης, να κάτσουν στο τραπέζι και να διαπραγματευθούν οι δύο πλευρές για να αποφευθούν τα χειρότερα. Γεγονός είναι ότι τα χειρότερα όμως αφορούν ε, και πλήττουν τους πολίτες και όχι τις ηγεσίε των δύο πλευρών, γιατί αυτοί οι οποίοι, ε, τους οποίους θα έπρεπε να αφορά η διαμεσολάβηση δεν συμμετέχουν σε αυτή. Η στασιμότητα ωστόσο υπάρχει και την έχουν διαγνώσει τα ΗΕ και γι' αυτό προσφέρουν τη διαμεσολάβησή του. Δυστυχώς αυτή η διαμεσολάβηση θεωρώ δεν είχε εξ αρχής πιθανότητες επιτυχίας, όχι μόνο γιατί διαμορφώθηκε όπως διαμορφώθηκε, γιατί ήταν αυτός που ήταν ο πρώτος διαμεσολαβητής, αλλά γιατί στη διεθνή κοινότητα είχε εκφραστεί μεν η ιδέα ότι ναι όλοι θα το στηρίξουμε, αλλά τελικά αυτό δεν υλοποιήθηκε. Πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές από τη διεθνή κοινότητα οι οποίοι έλαβαν, υποστήριξαν τη μία πλευρά ενώ ε, διακήρυταν την υποστήριξή τους για τη διαμεσολάβηση, όποιος ήταν ο διαμεσολαβητής, στην περίπτωση της Αιγύπτου και των Εμμυράτων υποστήριζαν τον Χάφταρ και τα στρατεύματά του. Ήδη δηλαδή ήταν μεροληπτική, μεροληπτική η ε, διαμεσολάβηση και δεν είχε ελπίδα επιτυχίας. Ήδη όμως, όπως είπα, εξ αρχής ο σχεδιασμός της ήταν ελαττωματικός, δεν είχε αρκετά ανοιχτή ε, όραση, δεν είχε σχεδιασμό δηλαδή που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιτυχία. Αλλά πρέπει και αυτό να το αντιληφθούμε ως ελάττωμα αυτής της διαμεσολάβησης. Και βέβαια φαίνει τις συνεπίες του και αυτό το ελάττωμα. Από εδώ και μπρος τι κάνουμε τώρα. Εάν παραμένει ο στόχος της διαφύλαξης, διάσωσης της μετάβασης σε ένα πλουραλιστικό σύστημα και άρα και της διάσωσης της ίδιας της Λιβύης, μπορούν να γίνουν τα εξής σε επίπεδο διεθνού κοινότητα, ασχέτω του τι θα γίνει στην ίδια τη χώρα, εμεί από τη δική μα την πλευρά, πώ μπορούμε να προβάλλουμε εξουσίε, υποστήριξη κτλ. Πρώτη επιλογή, προφανή, να αναζητηθεί, να εξευρεθεί μια πραγματική ενότητα ε, και ε, υποστήριξη της συμφιλίωσης ε, στην αποστολή Σαν Σαλαμέ, χάρη στην αποστολή Σαν Σαλαμέ. Αυτό είναι δεδηλωμένη βούληση. Και αυτό δηλώνει το ΕΕ Έθνη ότι είναι η μόνη λύση αυτή, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τι σημαίνει. Περιορίζονται μόνο στις εκηρύξεις. Μέχρι εκεί καλά. Ο στόχος ποιος είναι. Ο στόχος είναι η συμπαγής αντιμετώπιση, η υποστήριξη του Σαλαμέκ και εξασφάλιση τη δική του υποστήριξη για το σχέδιο συμφιλίωσης. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και το συζητήσαμε και στο παρελθόν. Ο Σαλαμέ σχεδίασε ένα σχέδιο το οποίο επί χάρτου έχει μια βάση, είναι εύστοχο, τροποποίηση της πολιτικής συμφωνίας, αλλαγή σε, από 9 σε 3 των μελών του Κυβερνητικού Συμβουλίου κτλ. κτλ. Μέχρι εκεί αυτή η ιδέα πάει καλά. Μετά πρόκειται να γίνει μια ε, εθνική συνέλευση, το δυνατόν πιο περιεκτική για συμπερίληψη των δυνατών τρών πλευρών, που θα οδηγούσαν σε συζήτηση όλε τι πλευρέ, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώ θα συζητούσαν. Αλλά, περιπτώσει, σημαντικά θέματα για το μέλλον της χώρας Και άρα θα προετοιμαζόταν με τον τρόπο αυτό ο δρόμος για τις εκλογές. Και μάλιστα και πριν από, τη σύνταξη, από την κατάρτιση συντάγματος θα γινόντουσαν εκλογέ. Αλλά δεν είχε εξηγήσει ο Σαλαμέ την αλληλουχία των δράσεων. Το προηγούμενο Σάββατο στην Ρώμη μάλιστα διευκρίνησε ότι δεν υπάρξει τροποποίηση της συμφωνίας του LPA και επειδή ακριβώ δεν υπάρχει συμφωνία γιατί οι δύο επιτροπές δεν έχουν συμφωνήσει, ούτω ή άλλω θα πάει στην Εθνική Συνέλευση. Στην Συνέλευση ναι. Και αυτό σκοπεύει να το πράξει Φεβρουάριο-Μάρτιο. Εσείς δεν ξέρω τι φρονείτε από αυτού, αλλά για μένα είναι σοβαρό πρόβλημα μια τέτοια επιλογή. Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει. Και μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για εκείνους που δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτρέψουν μια μετάβαση. Και έτσι μια στρατιωτική ομάδα ε, θα μπορούσε να αναλάβει τα ενία της χώρας, ακριβώς γιατί δεν έχει γίνει η μεταλλαγή της χώρας και γιατί μια τέτοια εθνική συνέλευση θα κρατούσε πάρα πολύ χρόνο. Λένε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και εδώ οι λεπτομέρειες είναι ο χρονισμός, η αλληλουχία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι με μια τέτοια πρόβλεψη μέχρι το Φεβρουάριο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μια δεύτερη εναλλακτική και εδώ παρακαλώ πολύ το λέω και θα σας παρακαλώ να το, να το αντιληφθείτε έτσι, το λέω ως πρόκληση μόνο για να προκαλέσω τη συζήτηση και όχι γιατί το πιστεύω. Εάν δεν αλλάξει το σχέδιο, αν, αν το σχέδιο Σαλαμέ δεν φέρει αποτελέσματα, αντί να κάτσουμε και να περιμένουμε το δεύτερο στάδιο, το δεύτερο βήμα, που θα ήταν ή ούτως ή άλλως οργάνωση μιας εθνικής ε, συνέλευσης, Α γίνει απευθεία η προκήρυξη των εκλογών. Αμέσω. Δύσκολο να οργανωθεί. Νόημα μπορεί να μην έχει γιατί δεν υπάρχει σύνταγμα. Είναι τόσο πολύ ιστορικά εκτοπισμένοι που θα είναι τεράστια η δυσκολία τη οργάνωση, τόσε δυσκολίε και τόσα προβλήματα και τόσε αντιρρήσει βέβαια μπορούν να διατυπωθούν ω προ την ιδέα τη εξαγωγή των εκλογών τώρα. Αλλά εάν το σχέδιο του Σαλαμέ δεν φέρει αποτέλεσμα, είναι η μόνη εναλλακτική αυτή που βλέπω να επανέλθουμε και να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο του πολιτικού γίγνεσθε. Πρέπει να τους απείσουμε τους πολίτες ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτές οι εκλογές και να αποφασίσουν οι πολίτες οι ίδιοι τι θέλουν, ποιος θέλουν να κυβερνήσει τη χώρα και με ποιους όρους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο μόνος τρόπος να κλείσουμε το δρόμο σε αυτούς που θα προτιμούσαν τη στρατιωτική αντιπαράθεση στη χώρα. Βεβαίως, αν επιλεγεί αυτός ο δρόμος έχει τεράστια σημασία ο ρόλος τον οποίο θα δερματίσει η διεθνή κοινότητα, κέρια σημασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να στηρίξουν αυτή την πορεία της Λιβύης προς τις εκλογές εγγυόμενες την παρατήρηση των εκλογών και την υποστήριξη της όλης διαδικασίας της εκλογικής. Και αν εξασφαλιστεί αυτό, πιστεύω, έχουν την ελπίδα οι πολίτες να ξαναγυρίσουν στο πολιτικό γείγναστο και να διασώσουν τη μετάβαση ίσως. Σταματώ εδώ. Και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω στο βαθμό που μπορώ τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαζάν. Ας ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σέντερ, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με το Μαγκρέμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Eh, Πραγματικά ήταν πάρα πολύ θετικό ε, οι παρεμβάσει αυτές, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τις ακούσω όλες. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει τεθεί το θέμα της διεύρυνσης της συμφωνίας και γύρω από την υπόθεση αυτή τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ήδη τέθηκαν από τους ομιλητές. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα από τα οποία προήλθε μια στήριξη στην προσπάθεια επίτευξης μιας πολιτικής συμφωνίας, μιας πολιτικής λύσης έτσι ώστε να ξεκινήσει επιτέλους μια εκλογική διαδικασία με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν βέβαια. Γνωρίζουμε το ιστορικό των εξελίξεων μέχρι σήμερα και έχουμε την αίσθηση ότι στην παρούσα φάση γίνεται μία απόπειρα γύρω από το κεντρικό θέμα της 16ης Δεκεμβρίου γίνεται μια προσπάθεια από τους διάφορους ε, πρωταγωνιστές τους οποίους ε, συναντήσαμε και μιλήσαμε. Υπάρχει λοιπόν μια απόπειρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα να υπάρξει ένα πριν και ένα μετά και να επιλεγεί ένας κοινός στόχος γύρω από αυτά τα οποία έχει ήδη πει όχι μόνο ο πρόεδρος Μακρό, αλλά και γενικότερα η διεθνής κοινότητα στα πλαίσια της έβρεσης των κατάλληλων συνθήκων που θα οδηγήσουν σε μια επαρκή εκλογική διαδικασία. Είχαμε λοιπόν συζητήσεις και συναντήσεις όχι μόνο με τον κύριο Σαλαμί, διαμορφώσαμε κάποιες απόψεις και θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε έτσι ώστε οι διάφορες πλευρές να θεωρήσουν ότι από τη στιγμή αυτή στα μέσα Δεκεμβρίου και μετά θα υπάρξει μια πλήρης επανεκκίνηση των διαδικασιών που θα βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν, να τα αγνοήσουμε αν θέλετε είναι αυτή η αίσθηση την οποία διαμορφώσαμε μετά από τις επαφές τις οποίες είχαμε, είναι προσωπική μου άποψη, συμπίπτει και με τις απόψεις ε, διαφόρων άλλων. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις ε, στα μεγάλα ερωτηματικά τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν κυρίως δε το πώς και τα ευρωπαϊκά όργανα και όσοι θέλουν να βοηθήσουν θα μπορέσουν σε επίπεδο συνεργασίας να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να είναι βαθιά πολιτική. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνει η διακοινοβουλευτική μου αντιπροσωπεία, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Ευχαριστώ. Περνάμε στις πολιτικές ομάδες. Δύο λεπτά η καθεμία παρακαλώ. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Γκάχλερ. Ναι, ευχαριστώ. για την παρουσίαση και τις θεωρήσεις σας. Ένα πολύ επίγον θέμα, πρακτικό, θα με απασχολήσει μόνο γιατί γνωρίζω λίγα πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και την Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης. Φαντάζομαι θα την παρακολουθήσατε κι εσείς όπου εκδηλώθηκαν πολλές καλές προθέσεις, έγιναν ωραίες ομιλίες ε, και παρουσιάστηκαν πολιτικές ε, ήδη υφιστάμενες, αλλά κάτι καινούριο στο πλαίσιο των συζητήσεων ήταν ότι εννέα κράτη συμφώνησαν ότι η κατάσταση αυτή των ε, καταβλισμών των προσφύγων είναι τόσο αποκαρδιωτική που θα πρέπει η Διεθνής Οργάνωση για τη Μετανάστευση να επιτρέψει είτε την ανάδειξη νέων καταβλισμών είτε να αναλάβει εκείνη τη διαχείριση των εφισταμένων και να επιτρέψει και τον επαναπατρισμό των προσφύγων αφενός αλλά και την ε, διαχείριση των ετοιμάτων, εκείνων που πραγματικά μπορούν να αποδείξουν ότι διώκονται πολιτικά. Μια περίπλοκη βέβαια απόπειρα, ένα περίπλοκο εγχείρημα. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω εσείς πώς αξιολογείτε αυτή την εξέλιξη γιατί βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν ε, πέραν των επίσημα αναγνωρισμένων καταβλισμών ε, προσφύγων και ιδιωτικές φυλακές όπου κρατούνται παράνομα ε, οι πρόσφυγες είτε για να ανταλλαχθούν με λίτρα είτε για να απολυθούν σε σκλαβοπάζαρα. Βλέπετε κάποια δυνατότητα να μπει ένα τέρμα σε αυτήν την αφόρητη πια κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν επιτρέπετε, έχω ένα πολύ λεπτομερές ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω στους ομιλητές. Γιατί λαμβάνουμε ιδιαίτερα γενικόλογες πληροφορίες για αυτό το αποτρόπαιο φαινόμενο με τη διακίνηση ανθρώπων από διακινητές που δεν έχουν ε, καμία δουλειά να κάνουν τέτοια πράγματα στη Μεσόγειο. Θα θέλαμε περισσότερες ε, πληροφορίες για το ποιος εμπλέκεται και με ποιον τρόπο υπάρχει στήριξη προς τα θύματα των διακινητών εάν εμπλέκεται ο στρατός, εάν υπάρχει τρόπος ε, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Οι δημόσιες αρχές ή ο στρατός κάνουν κάτι για να δώσουν ένα τέλος αυτή την ιστορία. Θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες λοιπόν ακριβώς για την διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Ευχαριστώ κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, αλλά έχω βραχνιάσει, ελπίζω να μην ε, δημιουργήσω πρόβλημα. Ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, για την κατάσταση των μεταναστών ήδη το έθιξαν ε, κάποιοι συνάδελφοι και αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος, όμως δεν υπάρχουν ε, επαρκείς πόροι. Συμμετέχουμε λοιπόν σε μία αποστολή που θα πάει στη Λιβύη. Ε, έπρεπε να είχε πάει μάλλον το Σεπτέμβριο, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν πήγε της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως βρήκαμε πολλούς ε, συνομιλητές στην Τίνιδα. Πρώτον, λοιπόν, πώς ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την ευρωπαϊκή συνδρομή σε αυτά τα ζητήματα. Η συμφωνία που υπήρξε υπό την ε, συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης, κατά πόσο μπορεί να τηρηθεί, τι γίνεται με την εκένωση εντός εγωγικών των μεταναστών πώς μπορεί να γίνει αυτή σε βάθος ε, έρευνα, καθώς ξέρουμε ότι και το δικαστικό σύστημα, η αστυνομία, ακόμα και ο στρατός, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ε, επίσημης κυβέρνησης, μπορούν να δράσουν μόνο σε ένα πολύ μικρό τμήμα της επικράτειας. Θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, για την κατάσταση στους καταβλισμούς. Του ανεπίσημου καταβλισμού όπω ανέφερε ο συνάδελφο προηγουμένω, που είναι και στην πλειοψηφία του, βέβαια τέτοιοι ανεπίσημοι. Είδαμε ε, και από τον και από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση μα είπαν ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί ένα καταβλισμό από επίσημο να γίνει ανεπίσημο. Γιατί έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Πώ γίνεται λοιπόν να ε, τηρηθούν αυτέ οι δεσμεύσει, ποιο μπορεί να αναλάβει αυτό το καθήκον ε, για να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντι στην διεθνή κοινότητα. Συνεχώς ε, προωθούμε το ζήτημα των ε, τοπικών αρχών. Και πράγματι πιστεύω ότι στη Λιβύη αυτό είναι μια πραγματικότητα, οι αρχές οι τοπικές. Οπότε και προς τους δύο. Πώς θεωρείτε ότι αυτές οι τοπικές αρχές μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα που ανέφερε ο καθηγητής, όσο γίνεται πιο περιληπτικό αυτό το εγχείρημα και αν τελικά οι τοπικές αρχές θα είναι αυτές που θα μας επιτρέψουν ε, αυτή την επανένωση και την βελτίωση των συνθηκών σε σχέση με σήμερα. Ευχαριστούμε. κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τα ερωτήματα μου είναι τα εξή. Πρώτον, για την κατάρτιση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Λιβική Ακτοφυλακή. Έχουμε πολλά ε, γεγονότα που είδαμε ότι υπήρχε παρεμπόδιση ε, επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών και στρατιωτικών σκαφών. Τι κάνετε εσείς ακριβώς για να διασφαλίσετε την παρακολούθηση των ακτοφυλακών μετά για τον βασανισμό, απαγωγή, πώληση και δημοπράτηση μεταναστών και προσφύγων. Ήδη τον Φεβρουάριο του 2016 είχαμε ψήφισμα του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα. Το Φεβρουάριο του 2016 συζητήσαμε με τον ε, Μάρτιν Κόμπλερ τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ και αυτό το ανέφερε. Το Γενάρη του 2017 η γερμανική πρεσβεία στον Νίγηρα μίλησε για ε, συνθήκες ε, στρατοπέδων συγκέντρωση σε συγκεκριμένου καταβλισμού και με τον Ιούνιο με τον κύριο Κούμπλε εξετάσαμε και πάλι τι ίδιε εκθέσει, τα ίδια ζητήματα και τώρα τον 15 Νοεμβρίου έγινε λόγο για σκλαβοπάζαρα. Και τώρα πρέπει να θέσω το εξή ερώτημα προς όλους. Τι σας εμποδίζει να σώζετε, σώσετε αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις ε, συνθήκες δουλείας. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά την ε, πλευρά της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Τόμπρουκ, γιατί δεν υιοθετεί το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ. Γίνεται λόγος για ένα νέο σύνταγμα, για παράδειγμα, ότι κανείς θα πρέπει να συμμετάσχει σε μελλοντική κυβέρνηση στη Λιβύη όποιος έχει νυφευθεί αλλοδαπό ή έχει διπλή υπηκότητα, διπλή ηθαγένεια. Αυτό πώς προκύπτει ακριβώ, τι κρύβεται πίσω από αυτό το αίτημα. Ξέρω μόνο από το Σύνταγμα ε, στη Μιανμάρ, όπου σκοπίμω ο στρατός δεν ήθελε η αν να έχει εξέχουσα θέση. Αλλά εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί σημαίνει αυτό. Και μετά έχουμε δύο εντάλματα σύλληψη κατά του Σάιφερ Καντάφη και ε, του πρώην επικεφαλής ε, της μυστικής υπηρεσίας. Ο Σάιφελ Καντάφη αφέθη ελεύθερος από τις πολιταφυλακές και ζει στη Λιβύη. Πώς ε, βλέπει το ρόλο του σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό και επίσης τι μπορεί να γίνει ε, για την υλοποίηση και την εκτέλεση αυτών των ενταλματών σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Ευχαριστώ κύριο Καστάλντο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Thank you, Σουκράν. Τρεις ερωτήσεις έχω. Η μία είναι σχετική με την ερώτηση της κυρίας Βερζιά. 120 εκατομμύρια δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Λιβύη και 182 εκατομμύρια για, για σχέδια για τη μετανάστευση, 162 για το καταπίστευμα για την Αφρική και 120 εκατομμύρια για διμερή βοήθεια και ακόμη 80 εκατομμύρια έχει διαθέσει η Ιταλική κυβέρνηση για να υποστηρίξει την ε, Λιβική ακτοφυλακή. Εσείς κύριε Φαρχάτη, είπατε ότι δεν είναι επαρκής στις συνθήκες ασφαλείας, το κάνει για τους ίδιους τους Λιβύους. Τα χρήματα αυτά πώς τα κρίνετε. Είναι σωστό να δαπανώνται αυτή τη στιγμή και με αυτόν τον τρόπο. Είναι πρόσφορο. Φτάνουν στον ε, στόχο τους. Βλέπετε κάποια πρόοδο ή αλλιώς βλέπετε κάποια, κάποιο τρόπο βελτίωση της κατάστασης ώστε να μην καταλήξουν στα λάθος χέρια τα χρήματα αυτά. Και δεύτερον, πιθανή αποστολή στη Λιβύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασφαλώς θα αποτελέσει και την ευκαιρία να εκδηλώσουμε την ε, αλληλεγγύη και την ε, υποστήριξή μας ε, και την προσήλωσή μας στον λαό της Λιβύης και την προσπάθεια να στηρίξουμε την πολιτική διαδικασία. Διερωτώ με όμως, τι μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια επίσκεψη, είναι κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια επίσκεψη. Και υπάρχει κίνδυνος ο Καλήφα Αφτάρ να προσπαθήσει να δράξει την ευκαιρία για να καταλάβει την εξουσία με την επίσκεψή μας ταυτόχρονα. Και επίσης για τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές ε, που αναφέρατε στο επόμενο νεάμινο Βεβαίως ε, πολλά μπορούν να συμβούν, θα μπορούσε και να καταληφθεί ο έλεγχος της ε, Τρίπολης. Από την άλλη όμως, όταν λέτε ότι πρέπει να γίνουν πρόορες εκλογές, πώς θα το εξασφαλίσουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε την ε, διαξαγωγή τους κατά τρόπο δημοκρατικό, χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο, πώς θα γίνει να συνδυαστούν με ένα νέο σύνταγμα και ο κύριος Ματόλτο, φίλος που δεν είναι εδώ τώρα, έχει πει ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο με συνταγματική νομιμότητα και ε, ανώθευτες εκλογές. Επομένως, πώς θα γίνουν εκλογές ανώθευτες και επιπλέον πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αμφισβητήσουν την επομένη των εκλογών ή χαμένη το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα Είμαι πολύ σύντομος, θέλω να καλωσορίσω τους ε, φιλοξενουμένους. Να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Φερχάτ. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι στάσεις τις οποίες στηρούν σημαντικές γειτονικές χώρες όπως η Αιγύπτος και η Αλγερία στη διαδικασία εξομάλυνσης και εκδημοκρατισμού της κατάστασης στη Λιβύη. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις για ένα θέμα το οποίο θεωρώ σημαντικό. Είναι δύο σημαντικοί περιφερειακοί εταίροι. Ε, ποιος είναι ο ρόλος τους στις εξελίξεις εσωτερικές στη Λιβύη. Λοιπόν δεν υπάρχει άλλος να θέσει ερωτήσεις, οπότε θα δώσω το λόγο για τις απαντήσεις. Δέκα λεπτά ο καθένας παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Στα εκλεκτά μέλη θα ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Γκάλα. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι τώρα για τον μηχανισμό ο οποίος έγινε αντικείμενο συμφωνίας της συνάντησης κορυφής ε, Αφρικανικής Ενότητας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αμπιτζάν περιλαμβάνει την πρόταση ο ION να διαχειριστεί ε, το κέντρο αφήξης ε, διαμετακόμισης και αναχώρησης στη Λιβύη να καλυφθούν έτσι οι ανάγκες επιστροφής των προσφύγων στις χώρες προέλευσής τους. Δεν έχει υπάρξει κάποια τεχνική τεκμηρίωση γύρω από το μηχανισμό αυτό και δεν μπορούμε πραγματικά να δούμε πού θα ε, έχει έδρα η υπηρεσία αυτή, στην Τρίπολη, εκτός Τρίπολης, στη Δυτική Λιβύη και οι αριθμοί οι οποίοι κυκλοφορούν ε, στο περιθώριο της συνάντησης του Αμπιτζάν είναι ότι θα ξεκινήσει με 3.700 ή 800 πρόσφυγες. Αυτός ίσως να είναι ο συναλλικός ε, αριθμός των προσφύγων σε ένα από τα κέντρα κράτησης, όπως το ονομάζουμε, στην Τριπολίτιδα. Από την πλευρά μας πάλι, από πλευρά της Λιβύης, ε, το ερώτημα το οποίο παραμένει είναι πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν όταν έχεις εκτοπισμένους, όταν έχεις απάτριδες, όταν έχεις πρόσφυγες. Είναι αδύνατο ε, τα Ηνωμένα Έθνη και η αρμοστία ε, να τους ε, βοηθήσει να επαναπατριστούν σαν παράδειγμα, έχουν έχουν καταγράψει μέχρι τώρα 43.000 απάτριδες και εκτοπισμένους. Αυτός είναι ένας αριθμός για τον οποίο εμείς στη Λιβύη δεν έχουμε ιδέα. Τον Αύγουστο του 2016 ο αριθμός αυτός υποτίθεται ότι ήταν 39.000 και ο αριθμός αυξάνεται έχετε τις, τα προγράμματα επανεγκατάστασης στην Ευρώπη. Προσπαθείτε να τα κάνετε να δουλέψουν, κατανέμετε τους πρόσφυγες με ποσοστώσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Ενώ εμείς στη Λιβύη δυστυχώς οι αριθμοί αυξάνονται και κανένας δεν μας λέει πότε θα σταματήσουν ε, να αυξάνονται και πότε θα περάσουν σε άλλες χώρες οι 47 αυτοί χιλιάδες πρόσφυγες και πολλοί πιστεύουν ότι άλλες 100.000 δικαιούνται ασύλου στη Λιβύη. Σύμφωνα λοιπόν και με την έκθεση του τέλους του 16 υπάρχουν συνολικά 700.000 πρόσφυγες συνολικά στο λιβικό έδαφος. Συνεπώς λοιπόν αν επανέλθω στον μηχανισμό που προβλέπεται για το κέντρο αυτό διαμετακόμισης και αναχώρησης το θέμα είναι πότε και πώς θα λειτουργήσει και πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες και πολλές από τις χώρες αυτές δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με τη Λιβύη. Ε, δεν είναι καν κοντά στη Λιβύη, οπότε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τις συνεννοήσεις που χρειάζεται. Και τι θα γίνει με τους κατοίκους της Ερυθρέα. Θα επιστρέψουν στην Ερυθρέα οι άνθρωποι αυτοί ή θα παραμείνουν στη Λιβύη. Όλα αυτά είναι εκκρεμότητες. Επαναλαμβάνω ότι 43 καταγεγραμμένοι, 43.000 καταγεγραμμένοι από τους μισούς, οι μισοί μάλλον είναι ε, Σύριοι και Ιρακινοί, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί από την Ερυθρέα, οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι καν καταγεγραμμένοι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα για μας και πρέπει να το αναφέρουμε. Εσείς εδώ στην Ευρώπη αποφασίσατε 20-22 επανεκαταστάσεις και έχετε εφαρμόσει μόνο 17-18 Με βάση την αρχή της επικουρικότητας έχετε δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής της απόφασης. Και είπατε ότι θα προχωρήσετε και με άλλους 50.000, κάτι το οποίο δεν είναι σαφές ότι θα πετύχετε πλήρως τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα για την σωματεμπορία και τη δουλεία εις βάρος των προσφύγων στην ε, Λιβύη. Κοιτάξτε, η πρακτική αυτή είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στη Λιβύη. Είναι κάτι το θλιβερό κάτι το οποίο απορρίπτει το σύνολο των Λιβύων, η Λιβική συνείδηση, η Λιβική κοινωνία. Δεν μπορεί ποτέ να αποδεχθεί αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες. Και αν υπάρχουν κάποιοι Λίβοι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί έμποροι Αφρικανοί οι οποίοι εμπορεύονται ανθρώπους και αυτό το κάνουν και σε λιβικό έδαφος. Η Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε την έκθεσή της για την δουλεία πέρυσι το Σεπτέμβριο, όχι μόνο στην Λιβύη όμως, αλλά από την Ιγυρία, από τον Νίγηρα. Υπάρχουν τέτοιου είδους πρακτικές μορφές δουλείας και σχετικά τώρα με την κατάσταση των ε, μεταναστών στα κέντρα κράτησης στη Λιβύη. η ορολογία κέντρα κράτησης δεν σας αρέσει. Εσείς θέλετε να τα ονομάσουμε κέντρα υποδοχής. Αλλά τα καταφύγια αυτά, ε, Γι' αυτά είναι υπεύθυνο το Υπουργείο, είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν 35 τέτοια κέντρα τα οποία διευθύνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Λέγεται ότι τώρα πια τα κέντρα αυτά φιλοξενούν 20.000 περίπου παράνομους μετανάστες, 20.000. Οι περισσότεροι από αυτούς συλλαμβάνονται στην θάλασσα και ε, επιστρέφονται σε 20 σημεία άφηξης των σκαφών με μετανάστες και μετά οδηγούνται στα κέντρα αυτά που ελέγχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάτι το οποίο πρέπει να προσθέσω σε σχέση με αυτό είναι ότι ο αριθμός των μεταναστών αυτών ισούται περίπου με τον αριθμό των Λιβύων πολιτών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πόλη της Ντάουαργα, δηλαδή είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Το κόστος εκπαίδευσης λοιπόν της ακτοφυλακής μας επιτρέπει να σώζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους επιστρέφουμε στην Λιβύη, αλλά δεν μπορούμε να φροντίσουμε τους δικούς μας πολίτες. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν και εσείς πώς έχει η κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν δεν θα πρέπει να βλέπετε ε, τη Λιβύη ε, σαν μια χώρα που ζει μια απλά χαόδης κατάσταση αποκλειστικά μόνο με το θέμα της μετανάστευσης. Είναι ένα πρώτο αν θέλετε τμήμα του ευρύτερου πακέτου αναγκών και απαιτήσεων για την Λιβύη, η οποία είναι μια χώρα που προέρχεται από πόλεμο και κανένα τα τελευταία 6-7 χρόνια δεν δίνει σημασία στην επικίνδυνη κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα μου. Και είναι περίεργο το οποίο ε, το να θέλει κανείς να λύσει τα προβλήματα μιας χώρας που βγήκε από τον πόλεμο μέσω της προστασίας μόνο των μεταναστών και μέσω της προστασίας απλά των μεταναστών από τις διεθνείς υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει λύση προς την κατεύθυνση αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν Η επίσκεψή σας είναι σημαντική. Θα πάτε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με Λιβύους θα επισκεφθείτε όχι μόνο τα κέντρα κράτησης, αναφέρθηκε και η κυρία Σέντερ, ε, θα επισκεφθείτε και τους Ταουργκάν οι οποίοι ζουν σε 17 στρατόπεδα γύρω από την Τριπολίτιδα και τη Βεγγάζη. Είναι γύρω στις 20 με 22 χιλιάδες από την πόλη της Ταούργα. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα στη χώρα μου. και στα πλαίσια τώρα της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση της ακτοφυλακής. Μετά από την δημιουργία του προγράμματος Σοφία, της επιχείρησης Σοφία, ξέρετε ότι η επιχείρηση αυτή είχε σαν μάχη την διάλυση των δικτύων σωματεμπόρων ουσιαστικά από το Μάιο του 2015 έως το Μάιο του 2016 κινητοποιήθηκαν όλα τα μέσα, λειτουργεί στα, α, στα εθνικά ύδατα της Λιβύης ε, το σύστημα. Από το 16 λοιπόν εκπαιδεύεται ε, η ακτοφυλακή για να αναλάβει την έρευνα και διάσωση ε, στις περιοχές που ελέγχονται από τη χώρα. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 150-160 που έχουν εκπαιδευτεί μέσα από τα σκάφη, μέσα στα σκάφη της Σοφία. Οι Ιταλικές αρχές έχουν δώσει τον Απρίλιο και τον Μάιο στην Λιβική Ακτοφυλακή τέσσερα σκάφη, τέσσερα ή πέντε σκάφη, όχι περισσότερα, Πριν από το Μάιο η ακτοφυλακή λειτουργούσε ε, μόνο ε, με ένα σκάφος όλο και όλο, 30 ε, μέτρων και που ήταν και ακατάλληλο για έρευνα και διάσωση. Τώρα λοιπόν με τα νέα σκάφη τα οποία μας διάφεσε η, η Ιταλία μπορούμε να παραμείνουμε στη θάλασσα σχεδόν 24 ώρες ακόμα και ε, με συνθήκες ε, ή μάλλον κυρίως όταν ε, οι συνθήκες είναι καλές. Από το Μάιο έχουμε αναχαιτήσει, ερευνήσει και διασώσει 17.000 πρόσφυγες, τους οποίους έχουμε επαναφέρει στην Λιβύη. Για τα προβλήματα τα οποία σημειώνουν οι ΜΚΟ, εδώ θα πρέπει να σας το εξηγήσω λίγο τεχνικά όταν τα σκάφη των παράνομων μεταναστών ε, δίνουν ένα σήμα στην ομάδα επαφής και αδιάσωσης στη Ρώμη, στέλνουν πολλές φορές την ίδια διακίνωση και στο σκάφος των ΜΚΟ που μπορεί να είναι η Μετσέν Sans ή η MOAS και αμέσως ε, στέλνεται ένα σήμα στην ακτοφυλακή όπου ε, λέγεται ότι υπάρχουν ορισμένα ελαφρά σκάφη στις συγκεκριμένες συντεταγμένες και πρέπει να βοηθήσετε στη διάσωσή τους. Οι ΜΚΟ όταν παίρνουν αυτή την ανακοίνωση προσπαθούν να φτάσουν νωρίτερα και να φτάσουν στα σκάφη με τους πρόσφυγες πριν φτάσουν τα σκάφη της Λιβικής Ακτιφυλακής και πριν ένα μήνα πάρα πολλοί έπεσαν στη θάλασσα από τους μετανάστες για να φτάσουν τα σκάφη των ΜΚΟ και όχι της ακτοφυλακής. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία ήταν περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα κύματα, θάλασσα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ε, δύσκολη, τα σκάφη αυτή είναι πολύ επικίνδυνη, τα σκάφη είναι μικρά και οι Αφρικανοί μετανάστες συνήθως δεν γνωρίζουν κολύμβηση και συμβαίνουν ανθρώπινες τραγωδίες και τελικά λοιπόν κατηγορείται η ακτοφυλακή της Λιβύης λες και από πρόθεση ήθελε να πνίξει τους μετανάστες αυτούς. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Η Λιβική ακτοφυλακή λειτουργεί υπό την ηγεσία Λίβιων αξιωματικών που έχουν πτυχία από στρατιωτικές σχολές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ελλάδας. Δεν είναι καλά καταρτισμένοι, αλλά τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους δεν είναι τα καλύτερα και τα σκάφη των Ιταλών δεν είναι και τα πλέον κατάλληλα για διάσωση γιατί για τη διάσωση χρειάζονται πολύ χαμηλά καταστρώματα από όπου μπορεί κανείς να πετάξει ένα δίχτυ ασφαλείας ή και με το χέρι να τραβήξει έξω να τους κολυμβητές μετανάστες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, συγκυρίες και τεχνικά στοιχεία που αφορούν αυτό το ζήτημα. Και θα μείνω εδώ να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μεζράν για να επανέλθω στα <laughs> υπόλοιπα στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ σημαντικά ερωτήματά σας. Σε ό,τι αφορά τη Συνόδο Κορυφή στην Αμπιτζάν δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Νομίζω ότι υπήρξε προσπάθεια βάσει αυτού του σκανδάλου με τα βίντεο, ε, τα σκλαβοπάζαρα από και από αφρικανικέ χώρε και από κάποιε ευρωπαϊκέ να πούνε εντάξει τώρα κάτι να κάνουμε. Όμως ε, πέραν στρατιωτικής επέμβασης τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει για τον πολύ απλό λόγο ότι εδώ και χρόνια λέμε ότι αγνοείται τι συμβαίνει στη Λιβύη, επιτρέπεται την κατα... καταρρεύση της δημόσιας τάξης, επιτρέπεται την παρίσφρηση των ε, παράνομων οργανώσεων, το άνοιγμα των συνόρων. Έχουν ε, πέρασει τα σύνορα άνθρωποι που, που δεν είναι λιβικής καταγωγής, οπότε να λέμε τώρα στην κυβέρνηση Σεράζ ε, ότι δεν κάνατε κάτι ενώ για χρόνια την αγνοούσαμε, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Και συμφωνώ με τα όσα ανέφερε ο κύριος Φαρχάτ. Ένα ερώτημα αφορούσε τις ε, τοπικές αρχές. Κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό είναι να επιλύσουμε το ζήτημα σε εθνικό επίπεδο πολύ απλά γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, σε τοπικό επίπεδο. Και ε, ουσιαστικά πρόκειται για μικρά πράγματα τα οποία λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις. Δεν λέμε ότι ε, είμαστε αντίπαλοι επειδή μου κλέψε πέντε πρόβατα ή μου κάνει κάποιο άλλο κακό, αλλά επειδή είσαι Ισλαμιστής ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει λοιπόν, αν λύσουμε την πόλωση, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και διαμεσολάβηση επιτόπου. Δεν πρόκειται να επανέλθει η μου κανει καποιο αλλο κακο αλλα επειδη εισαι ισλαμιστη η οτιδηποτε αλλο υπαρχει λοιπον αν λυσουμε την πολωση τοτε θα μπορεσουμε να εχουμε και διαμεσολαβηση επιτοπου δεν προκειται να επανελθει η λιβυη στο, σε ένα κεντρικό καθεστω οπω ήταν υπό τον Καντάφη. Πότε πρόκειται να επανέλθουμε εκεί. Χρειαζόμαστε ένα επικεντρωμένο σύστημα στο πλαίσιο βέβαια ενός ενιαίου κράτους, ε, με κατανομή πόρων, βάση για να υπάρχει και αναδιανομή του πλούτου σε τοπικό επίπεδο και ορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες και σε τοπικό επίπεδο. Όμως, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν μπορούμε να πάμε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Γιατί στη Λιβύη υπάρχει, υπάρχουν πολλά επίπεδα είναι ο τοπικός κυβερνήτης, ένα τοπικό συμβούλιο, υπάρχει άλλο δημοτικό συμβούλιο το οποίο δεν εκλέγεται τοπικά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνηση, Κάποιοι ε, κάνουν καλή δουλειά, κάποιοι άλλοι όχι. Όμω, ε, δεν είναι επανάκια απλώ να πούμε ότι εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο. Δεν γίνεται αυτό αυτομάτω. γιατί αναφέρεται στο προσχέδιο του συντάγματος ότι αν κάποιος έχει διπλή ηθαγένεια δεν μπορεί, να, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε και το καθεξής. Αυτό οφείλεται στην πολιτική απομόνωση, αν δεν κάνω λάθος. Όλη αυτή η ιδέα ότι, που προώθησαν οι Ισλαμιστές για να προωθήσουν ορισμένα πρόσωπα. Είμαι βέβαιος ότι σε μια αναθεώρηση ε, του συντάγματος ε, αυτή η διάταξη θα αφαιρεθεί. Ε, παρουσιάζεται λοιπόν και ως ε, πρόταση την εκτελεστική εξουσία. Το πιο σημαντικό είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Ε, συμφωνώ με το πώς το έθιξε ο Σελαμέ. Είπε ότι εμείς δεν μεροληπτούμε έναντι κανενός. δεν θα πούμε σε κανέναν ότι εντάξει δεν μπορείτε να κατεβείτε στις εκλογές. Πρέπει να υπάρξει πρώτα η επίλυση του ζητήματος ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και μετά να μπορεί κανείς ε, να εκλεγεί. Είτε να πάει σε δίκη είτε να υπάρξει κάποια άλλη λύση. Μετά κανένας δεν θα έχει πρόβλημα με, την, με συγκεκριμένες υποψηφιότητες όταν λυθούν αυτά τα ζητήματα. Κανεί στη Λιβύη δεν είπε όχι σε καμία περίπτωση. Αν θέλει, α κατέβει ποιο θέλει τι εκλογέ και βλέπουμε. Το πολιτικό ζήτημα είναι διαφορετικό. Μπορεί όντω να αποτελέσει ε, προσωπικότητα που θα ενώσει τη χώρα. Τώρα εκεί είναι θέμα προσωπικής γνώμης. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι, εκπροσωπεί ε, κάτι το αρνητικό και δεν θέλουμε να επανέλθουμε εκεί. Ε, όπως η Ιταλία μετά τον φασισμό απαγόρευσε την σύσταση τέτοιου κόμματος για να μην επανέλθει. Κάτι αντίστοιχο είναι ε, το να πει κάποιος ότι όχι δεν θα σας επιτρέψουμε να κατεβείτε τις εκλογές γιατί δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό το καθεστώς. Για τις εκλογές τώρα από τεχνική σκοπιά δεν είναι πρόβλημα νομιμότητας, αλλά νομιμοποίηση. Από νομική άποψη, εντάξει, μπορεί κάτι τέτοιο να διασφαλιστεί. Ο πρόεδρο ε, της Επιτροπή είπε ότι μπορεί να γίνει. Το πρόβλημα είναι πώ θα γίνει, ούτω ώστε η πλειονότητα των ε, Λιβιών να συμμετάσχουν για να νομιμοποιηθούν αυτές οι εκλογέ και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του 2014 που μόνο 15% πήγε να ψηφίσει. Αυτό είναι στρατηγική σημασία λοιπόν για τις εκλογές, εάν θα νομοποιηθεί ε, στα μάτια των πολιτών αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σε όλα τα στάδια και από τον εκλογικό νόμο, όχι σαν αυτόν του 12 που, που ήταν ιδιαίτερα περίπλοκος και κανείς δεν τον καταλάβαινε, αν έχουμε έναν απλό εκλογικό νόμο και έναν μηχανισμό εκστρατείας, εκλογικής εκστρατείας, να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πολύ σημαντική αναμέτρηση, τότε διασφαλίζεται και η νομοποίηση της εκλογικής αναμέτρησης. Σε αντίθετη περίπτωση καταλαβαίνω ότι αν δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει ε, και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν δεν υπάρχει αναλλακτική, Εάν δεν λειτουργήσει το σχέδιο Σαλαμέ, τότε από το να καθόμαστε στα τα χέρια, καλύτερα να απευθύνουμε μια έκκληση και να δούμε τι θα γίνει. Αν υπάρχει ισχυρή συμμετοχή στις εκλογές ε, και τοποθετηθεί ο λαός, τότε θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε ε, να αντιταχθεί σε αυτό. Ε, μπορεί να είμαι αφελής, αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι θα προλάβουμε τα χειρότερα για την ε, επίσκεψη των Ευρωβουλευτών. Είναι πολύ σημαντική. Όμως, ε, σας συνιστώ να μην το κάνετε γύρω στις 17 Δεκεμβρίου. Εγώ, στη θέση σας, θα την ανακοίνωνα σήμερα και θα έλεγα θα έρθουμε στις 10 Ιανουαρίου, κάπου εκεί. για να δούμε, να μην έρθουμε ακριβώς τη στιγμή ε, που θα γίνει όλη αυτή η συζήτηση. Αλλά θα έρθουμε κάποια στιγμή να ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται. Το Γενάριο όμως ή αργότερα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό εσείς. σχέση με τους βασανισμούς και απαγωγές εις βάρος μεταναστών στη Λιβύη. Οι απαγωγές δεν περιορίζονται μόνο στους μετανάστες. Και οι Λιβύοι πέφτουν θύματα απαγωγών για λίτρα. Και δολοφονιών ακόμη. Για το 2017 μόνο, ε, από την οικογένεια Σαρσάρη της Δυτικής Λιβύης, ένας πατέρας μας καταγγέλει ότι τα τρία του παιδιά είναι εδώ και τέσσερα χρόνια κρατούμενα, θύματα απαγωγής, δεν μπορεί να τα ε, ξαναφέρει πίσω στην οικογένεια, ούτε οι αρχές της Λιβύης. Και κάτι ακόμη για την ακτοφυλακή της Λιβύης και το σκάφος Ερκεφάχ που κάνει διάσωση. Ο καπετάνιος του πλοίου έχει γιο 14 ετών που προσπάθησε μια συμμορία να απαγάγει και όταν το παιδί προσπάθησε να ξεφύγει, τον πυροβόλησαν στο πόδι. Τώρα είναι ανάπηρο το παιδί, επειδή ο πατέρας του εργάζεται σε αυτό το σκάφος της διάσωσης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Είναι λίγα αυτά τα παραδείγματα, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τέτοια. Καλώ λέει ο Πρόεδρος. Δύο τελικά συμπεράσματα, ευχαριστώντα σα βέβαια για την παρουσία σα. εδώ. Πρώτο συμπέρασμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πιστεύω να με πιο πολύ σαφήνεια την κατάσταση, είδαμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, για συζήτηση της Λιβύης, του Λιβυκού προβλήματος και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα πρέπει πιστεύω να συζητήσει το θέμα αυτό αλλά και να φροντίσουμε να έχουμε μια ε, ενιαία στάση και τοποθέτηση, να μην λέει κάθε Επιτροπή τα δικά της, για να συμβάλλουμε και στη συζήτηση, για να μπορέσουμε να φέρουμε κάποια αλλαγή στο βαθμό που μπορούμε σε αυτή την ε, κατάσταση. Επί της ουσίας, γνωρίζουν πιστεύω οι προσκεκλημένοι μας, ότι η καταπολέμηση των ε, προβλημάτων στη Λιβύη θα εξαρτηθεί και από τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η επικάλυψη διαφόρων επιπέδων εξουσίας και αντιπαράθεσης μεταξύ αντίπαλων φατριών. Όντως η έκρηξη της βίας εμφανίστηκε το 2014 με τον ε, Αφτάρ και το Λιβικό στρατό αφετέρου, τις πολιτοφυλακές ε, στην περιοχή της Τρυπόλιδος το Μεζουράτα αλλά και άλλες περιοχές που δραστηριοποιήθηκαν οι πολιτοφυλακές. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση και βία που δεν επέτρεψε την συζήτηση και άλλο μεταξύ των διαφορών ε, πρωταγωνιστών. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της Λιβύης είναι πάνω απ' όλα υπόθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Η Λιβύη βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ε, έχει στρατηγική θέση για την στρατηγική και τη σταθερότητα, αλλά και γιατί είναι στο σταυροδρόμι των μεταναστευτικών ροών και ταυτόχρονα επειδή έχει τεράστια επίδραση η θέση της Λιβύης για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε σε μια ευρύτερη θεώρηση την ε, κατάσταση, την ε, σκακέρα και τους διάφορους παράγοντες η δική μας στάση πρέπει να αναπτυχθεί μέσα από μια στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που βεβαίως και συστήθηκε στην Επιτζάν, αναπτυξιακή πολιτική, μεταναστευτική πολιτική, ε, οικονομική πόρη που θα στηρίξουν αποτελεσματικά αυτές τις πολιτικές. Μετά χρειάζεται μια διαδικασία πολιτικής σταθεροποίησης Η πρόταση για τη διεξαγωγή εκλογών ε, του Σαλαμέ μπορεί να είναι ένα θέμα που μπορεί κανείς να συζητήσει, αλλά δεν πρέπει να προχωρήσει γιατί έχει ε, και εμπεριέχει άλλους παραγόντες κινδύνου που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και πιστεύω ότι πρέπει σήμερα να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια ώστε η συμφωνία της Κυράτ να διατηρηθεί και να παραταθεί και μετά τις 17, να μην είναι δηλαδή η 17η Δεκεμβρίου μια καταληκτική προθεσμία. Δεν έχει συμβολική σημασία, είναι σημαντική μεν ημερομηνία η 17η, αλλά πρέπει να δώσει στις διάφορες πλευρές την, ε, το περιθώριο το χρονικό για να χτίσουν μια διαδικασία συμφιλίωσης. Και βέβαια περιμένω και ανησυχώ ως προς την απάντηση που θα δώσει ο στρατηγό Σαφτάρ αλλά και γενικά ε, τάσεις ε, απόλυτες και βίες που μπορεί να επηρεάσουν την διαδικασία. Και κλείνω αναφερόμενο σε δύο τελευταίες πτυχές. Το μεταναστευτικό είναι τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνει διόρθωση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι χώρες, η δική μου η πατρίδα η Ιταλία, σπέβδουν και ε, αγωνιούν να κάνουν συμφωνίες, να συνάψουν συμφωνίες για να περιορίσουν το μεταναστευτικό βάρος που είναι τεράστιο για την Ιταλία. Συγκεκριμένα από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να ε, ισχυριστούμε ότι δεν βλέπουμε πω η απόθεση ε, δημιουργεί στην Λιβύη τεράστια προβλήματα. Αλλά όχι μόνο αυτό, και αυτό βέβαια πρέπει να το έχουμε υπόψη πάντα, αλλά ταυτόχρονα και ε, το ότι τα γεγονότα αυτή τη στιγμή και το ότι έχει ε, αποτύχει, έχει καταδικαστεί από τη στάση αυτή σε αποτυχία η προσπάθεια των λαθροδιακινητών, τους έχει φέρει τους έχει υποχρεώσει να περάσουν σε μια άλλη δραστηριότητα, δηλαδή τα σκλαβοπάζαρα και το λαθρεμπόριο του πετρελαίου. Και εδώ μιλούμε για σκάφη που μεταφέρουν πετρέλαιο και εδώ υπάρχει κίνδυνο συμφωνίες διμερείς απόθεσης να φέρουν δύο συνέπειες, αφενός μεν να εγκαταλειφθούν σε πολύ δύσκολες απάνθρωπες συνθήκες οι μετανάστες και η άλλη πτυχή είναι να προκληθεί μια προσαρμογή των δραστηριοτήτων των λαθροδιακινητών σε νέες ε, εγκληματικές δραστηριότητες που θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στη Λιβύη. Γι' αυτό χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση. Αυτό λέω και θα πω και στην έκθεσή μου. Και από όλη τη συζήτηση αυτή δεν μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση χωρίς να πούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο προς τους Υπάρχουν τεράστια περιφερειακά συμφέροντα εκτός της ίδιας της Λιβύης αλλά και της ευρύτερη περιφερειές της. Υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλες χώρες, οι οποίες πώς να το πω, έχουν με τι άλλο αμφίσιμη στάση και ως εκ του δεν επιτρέπουν την εξέβρεση μιας ε, κατάλληλη ισχυρή και ενωμένη αντίδραση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το οποίο θα πρέπει να θέσουμε ως ζητούμενο είναι μια σαφής εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική ώστε να δοθούν απαντήσει στο θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι καθήκον μας στη σύνταξη της έκθεσης για τη Λιβύη θα είναι να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα και να φροντίσουμε ώστε η ε, δημοκρατική σταθεροποίηση να βρει χώρο για να σταθεί, να εδρεωθεί και να αναπτυχθεί. Και βεβαίω ε, το θέμα αυτό ενδιαφέρει και τι άλλε επιτροπέ. Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα και συνθετική ε, στάση και ενωμένη παρέμβαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα και για τη διάθεση συζήτηση και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τη σημερινής διάταξη. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Συνεχίζουμε συνάδελφε με το δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μακροοικονομική βοήθεια προς την Γεωργία. Έχει ξεκινήσει μια σημαντική συζήτηση όπως γνωρίζετε, εμεί έχουμε θέσει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αιρεσιμότητα και σχετικά με την χρήση των πόρων οι οποίοι ε, έχουν σημειωθεί προς τη Γεωργία. Η συγητής είναι ο κύριος Μαμίκης, στον οποίο δίνει το λόγο αμέσως. Thank you, Chair. As you have... Όπως είπατε, Πρόεδρε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δώσουμε 45 εκατομμύρια στην Γεωργία σε επίπεδο δανείων και δωρεάν βοήθεια τα υπόλοιπα. Η τελευταία πληρωμή έγινε τον Μάιο του 2017. Οι άλλες χώρες στα πλαίσια του ιδίου προγράμματος είναι η Τινησία, ο Λίβανος, η Κυργιζία, η Ιορδανία, η Ουκρανία και η Γεωργία. Υπάρχει μία τροπολογία στα πλαίσια της κοινή δήλωσης. Στόχος είναι να επιβεβαιωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ε, μακροοικονομικής ε, συνδρομής ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Δεύτερον, να είμαστε σίγουροι ότι η υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων θα παρακολουθήσει την πλήρη λειτουργία του προγράμματος καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και τέλος να διασφαλίσουμε την ε, συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γύρω από αυτό. Η αιρεσιμότητα στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής θα βοηθήσει να δοθούν κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της δημοκρατίας και στον τομέα του κράτους δικαίου. Το κράτος στη Γεωργία προσπαθεί να προωθήσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σύμφωνα και με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να προσθέσω εγώ ότι η κοινή δήλωση ήταν μια λύση στην οποία είχαμε καταλήξει και για τη Μολδαβία τον προηγούμενο Μάιο. Αυτή τη φορά η διατύπωση που προτείνω είναι πιο θετική γιατί η Γεωργία αποδέχεται το σύνολο των συστάσεων της Βενετίας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις λεπτομερέστατες απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Τα έλεγξα τα θέματα αυτά με τους σκιώδεις συναδέλφους και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους. Να ευχαριστήσω επίσης και τον γνωστό συνάδελφο Τάκουλα, και η δική μας Επιτροπή και η ΙΝΤΑ συνεργάζονται για να προωθηθεί η υπόθεση αυτή το ταχύτερο δυνατόν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή. Εκτιμώ ε, τη συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών μας και ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τον εισηγητή. Ήταν πολύ αγαστή συνεργασία μας. Με τα χαράς να ακούσω και τα δικά σας ε, σχόλια στη συνέχεια. Είναι η τρίτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ε, μακροοικονομική αρρωγή προς τη Γεωργία μετά την ε, στρατιωτική διένεξη με τη Ρωσία το 2008. Αυτή τη φορά προτείνεται αρρωγή ύψου 45 εκατομμυρίων. Τα 10 θα δοθούν μέσω ε, επιδοτήσεων και τα υπόλοιπα 35 μέσω δανείων. Η Γεωργία είναι χώρα της ανατολικής τερικής σχέσης με ε, δύσκολη γεωπολιτική θέση. Τα τελευταία χρόνια το νόμισμα έχει υποτιμηθεί σημαντικά και αυτό έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη του ε, χρέους. Η οικονομία έχει πέσει εξαιτία των ε, μειωμένων εξαγωγών, εμπορικών εξαγωγών και το, το ΑΕΠ διατηρείται στα επίπεδα του χάρη σε επενδύσεις. Διατηρούνται όμως κάποια ε, επίπεδα στο χρηματοοικονομικό επίπεδο ε, χάρη στην επίβλεψη από την Κεντρική Τράπεζα. Πρόσφατα έχει συναυθεί και, ε, και Συμφωνία των λαγών το οποίο επιτρέπει τη σταθεροποίηση της γεωργιανής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει συστάσεις στη Γεωργία για το πώς να προχωρήσει στην δημοκρατική σταθεροποίηση αυτή η διαδικασία βέβαια παίρνει χρόνο. Και προκειμένου να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις ε, θα πρέπει να βασιστούμε σε μέτρα που θα ληφθούν από την ίδια τη χώρα. Θεωρώ ότι η Γεωργία έχει αποδείξει την βούλησή της ε, να συνεχίσει να κατευθύνεται στον δρόμο της ε, σταθεροποίησης και η δική μας αρρωγή θα βασίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την πρόοδο που σημειώνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρέντα ε, που αντικαθιστά τον ε, κύριο Στέτινα. Ευχαριστώ πολύ. Παίρνω το λόγο εξ ονόματος ε, του συναδελφού Στέτινα, που είναι σκιώδης συγητής μας. Πρώτον, ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους για την πρόταση επί της διαδικασίας ο κύριος Στέτινα συμφωνεί με τα όσα προτείνει ο κύριος Μαμένκινς, δηλαδή υποβολή τροπολογίας ε, με τη μορφή ενιαίας ε, δήλωσης ε, των τριών θεσμικών οργάνων. Γνωρίζουμε ότι η Γεωργία τα πηγαίνει πολύ καλά, όμως πάλι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. ο κύριος Στέτινα αναφέρει ιδίω βάσει της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε υποθέσεις για τη σταγματική αναθεώρηση. Σε ό,τι αφορά την ε, μακροοικονομική διαχείριση και την ε, λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και με την αμερόληπτη δικαιοσύνη, όλα αυτά πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στην κοινή μα διακήρυξη. Όμω θα πρέπει να ελοπιθεί και στην πράξη. Βάσει του άρθρου 12 της πρότασης της Επιτροπής, ε, η Επιτροπή και οι Δράσεις θα παρακολουθούν την προϋπόθεση για την χορήγηση της ενωσιακής μακροοικονομικής αρρωγής όλο τον κύκλο ζωής του. Το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι αυτές οι προϋποθέσεις είναι ο σεβασμός προς ε, τους ε, δημοκρατικούς θεσμούς, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να διευκρινίσουμε τη διαδικασία, λέει ο κ. Στέτινα, έχω ένα ερώτημα προς ε, τον εκπρόσωπο των δύο αυτών θεσμικών οργάνων της Επιτροπής και της Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης, που θα εποπτεύουν τη διαδικασία αυτή. Το πρώτο ερώτημα που απευθύνει ο κ. Στέτινα είναι το εξή. Μπορείτε παρακαλώ να περιγράψετε λεπτομερώς πώς ε, η αιρεσιμότητα που περιγράφεται στο άρθρο 2 θα υλοποιηθεί και δεύτερον, η κοινή μας ε, διακήρυξη είναι ένα εργαλείο μόχλευσης για, για να δώσουμε κίνητρο για την ε, εκδημοκράτηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Και ο κύριο Σίτιν επίση προσβλέπει στη συνεργασία με τον εισηγητή και άλλου κοιότε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαστρεβίτσιου. Ευχαριστώ συνάδελφοι που δίνει τη δυνατότητα να σας ε, μιλήσω για αυτό το ζήτημα εξ ονόματος του Χαβιά Νάρθα, του συναδέλφου που είναι σκιώδης από πλευρά Σάλντε. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι είναι σημαντική η στιγμή εφόσον όλα είναι και περισσότερο δίνουμε έμφαση στις επιδόσεις και στην ε, υλοποίηση των συμφωνιών σύνδεσης καθώς και των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών με τις ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστή πολιτική κατεύθυνση. Ε, είναι σωστή και η απόφαση της ΑΦΕΤ ε, να έχουμε εκθέσεις προόδου του χρόνου για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις για αυτές τις χώρες δηλαδή που είναι διατεθειμένες να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές από τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πράγματι, είναι σωστή η αιρεσιμότητα εδώ. Ακόμα και αυτή η τροπολογία που με κάποιον τρόπο συνδέει πολιτικά κριτήρια με την μακροοικονομική αρρωγή. Έχει έρθει η ώρα, συνάδελφοι, να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτής της, ε, αυτού του συσχετισμού, όχι για να τιμωρήσουμε κανέναν, απλώς ε, για να θεσπίσουμε ένα σημαντικό μέσο παρακολούθησης και επιρροής η άσκηση της επιρροής ε, στην κατάσταση σε ορισμένες χώρες. Διαφέρει λοιπόν η δημοσιονομική και η μακροοικονομική στήριξη. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και νομίζω ότι υπήρξε μια συμφωνία τελικά μεταξύ των όσων συμμετείχαν στη συζήτηση. Και εφόσον έχουμε την ίδια τροπολογία και την ίδια κοινή δήλωση για τη Μολδαβία, θεωρώ απόλυτος ε, σκόπιμο να γίνει το ίδιο και με τη Γεωργία. Και συνάδελφοι, συμφωνούμε ότι όλα αυτά που εξετάζουμε θα πρέπει να ε, βαίνουν υπέρ των χωρών αυτών σε ό,τι αφορά τον κώδικα διοντολογίας, τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αυτές τις χώρες, σε ό,τι αφορά την χρήση και αξιοποίηση της στήριξης που παρέχουμε ορθά σε αυτές τις χώρες. Και ο συνάδελφος Χάνου Τάκουλα θα μας ε, στηρίξει σε αυτήν την πολιτική σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό συνέδριο και έτσι θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όσον αφορά την τελευταία επιθυμία του συναδελφού Αστρουίτσους, δεν μπορώ παρά να την υποστηρίξω. Κύριε Στάκουλα, Έμαθε πολλά από την Ίντα. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια τον εισηγητή για το σχέδιο στην Ίντα. Είχαμε μια εισβάθος συζήτηση για τη στόχευση και τις, μακρο... και τις θετικές το θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει μακροοικονομική υποστήριξη, αλλά βέβαια και προβλήματα μπορεί να γεννηθούν σχετικά. Και δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω και να ε, τονίσω τη σημασία της αιρεσιμότητας ως μέσου και τα όσα έχει να πει βέβαια και η ΑΦΕΤ για τις χώρες της εταιρικής σχέσης. Αυτό σημαίνει, ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς τη διαδικασία, όχι μόνο με εκθέσεις ε, μια φορά το χρόνο. Όλες οι δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή την ε, ε, παρακολούθηση γιατί δίνουμε τα λεφτά του ε, Ευρωπαίου φορολογούμενου και εμείς είμαστε υπόλογοι μετά να εξηγήσουμε στον πολίτη αυτά τα χρήματα ε, που πήγανε. Και κάτι ακόμη που σχετίζεται με μια πιο συγκεκριμένη αναγνώριση και αναγνωρισμότητα του πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά στους εταίρους μας εν προκειμένου τη γεωργία. Εξού και η τροπολογία για τα νομικά ζητήματα. Συστάσεις της Επιτροπής Βενετίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά ταυτόχρονα εδώ στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να συμπληρώσω και με ένα επιπλέον στοιχείο ότι πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των δανείων και των δωρεών. Ε, τα δάνεια πολλές φορές επαναλαμβάνεται ότι μπορεί να ε, κρατήσουν μέσα σε ένα ε, κύκλο εξάρτησης τα κράτη αυτά από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να χτίσουν τις οικονομίες τους, να τις στηρίξουν όπως εννοούν τα ίδια με, το δημοκρατικό, με τη δημοκρατική επιλογή όλων των ε, κατοίκων τους ώστε να σταθούν αυτόνομες οι οικονομίες των κρατών αυτών και γι' αυτό για την ομάδα μου είναι προτιμότερες οι δωρεές από τα δάνεια γιατί έτσι πραγματικά τους δίνουμε πρόσθετη οικονομική υποστήριξη να την διαθέσουν όπως θεωρούν σκοπιμότερο. Ευχαριστώ. Thank you. So, um, I... Η κυρία Χάρμς, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη συζητήσει σε μια σύνοδο κορυφής για τις χώρες της Ανατολικής γειτονίας, και την Ανατολική γειτονία γενικότερα ε, τα ότι έπεται σε σχέση κυρίως με τις συνδεδεμένες χώρες και αν θα είναι περισσότερα ή λιγότερα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Όλοι συμφωνούμε ότι το επόμενο βήμα είναι πάνω απ' όλα η υλοποίηση των συμφωνιών σύνδεσης και αυτό που πρέπει να επιτύχουμε με τη μακροοικονομική ε, υποστήριξη, ενίσχυση είναι πάνω απ' όλα να δώσουμε έναυσμα για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται χάρη σε αυτή την υποστήριξη και, με τις, ε, και από τις συναντήσεις που είχαμε με τους εταίρους, συνδεδεμένες χώρες, εταίρους από και για τη γειτονία γενικότερα, ε, βλέπουμε ότι είναι αποδεκτή αυτή η λύση πολύ θετικά. Συμπληρώνω επίσης για τους συναδέλφους της ΣΥΝΤΑ την ιδέα ότι θα πρέπει να συζητηθεί και η δική μας αξιοπιστία ως προς τους όρους που ορίζουμε. Εάν δηλαδή ορίζουμε ε, όρους εφικτούς, πρέπει και να τους στηρούμε. Η διαδικασία του προσδιορισμού των όρων είναι για μένα ακόμη εκκρεμής, δεν έχει ολοκληρωθεί και για τους συναδέλφους της Euronest και τη συνεργασία με τις χώρες Ανατολικής Γειτονίας θα ήθελα να προσφέρω αυτή τη διάσταση για να την εξετάσουν. Για τη Γεωργία όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για μια χώρα που έχει πολύ καλύτερη ανάπτυξη από ότι άλλες αντίστοιχες χώρες. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές πιέσεις, γιατί έχουν όχι μόνο αυτές τις λεγόμενες παγωμένες συγκρούσεις, ε, ε, αλλά και το Αζερβαϊτζάν και την ε, Τουρκία, που φαίνεται να είναι πολύ διεκδικητική και γενικά οι γειτονικέ χώρες ασκούν πίεση. Άρα λοιπόν έχουμε πολιτική ένταση την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε κατά την αξιολόγηση μιας χώρας. Από ό,τι βλέπω εγώ και ύστερα από όσα είπατε, θα ήθελα να ε, συμπληρωθεί στην εξέταση και η εξέλιξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η διαφάνεια στον τομέα των ΜΜΕ, αλλά και τα ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτας καθεστώτος του ΜΜΕ και βέβαια του πλουραλισμού στα ΜΜΕ. Αυτά πρέπει να μπουν ως όροι ως αιρεσιμότητα, όπως και η ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Ήταν ένα από τα θέματα που επισήμαναν στη συζήτηση και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής της Βενετίας. Η ανεξαρτησία της ε, δικαστικής εξουσίας δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Έχουμε διαπιστώσει όντω θετικές εξελίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε με όρους ξεκάθαρους ε, τα θέματα αυτά με την εταίρο μας συνδεδεμένη χώρα Γεωργία. Και επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου ολοκληρώνοντας, διότι η Γεωργία είναι από τις λίγες χώρες που δεν ε, παραδίδει στην Τουρκία λεγόμενα μέλη του κινήματος Γκυλέν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και, και τη γνωρίζουμε ότι δεν αντιμετωπίζονται με τον ιδεώδη τρόπο πάντοτε όλα τα θέματα των ανθρωπών δικαιωμάτων και μάλιστα ζητήματα όπως αυτά των φύλων μάλλον με τρόπο κακό αντιμετωπίζονται, πρέπει και αυτό να υπολογιστεί μέσα στη γενικότερη στρατηγική και γεωγραφική θέση της Γεωργίας. Ευχαριστώ. Γιουρέκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό για μας να δοθεί υποστήριξη στη γεωργία για διάφορους λόγους για τη γεωπολιτική της καταρχάς θέση, για λόγους ιστορικούς βεβαίως, αλλά και άλλους αντικειμενικούς όρους, αλλά και για λόγους ε, υποκειμενικούς. Η κοινωνία της γεωργίας θέλει να έρθει πιο κοντά στις δυτικές χώρες. Συμφωνώ πάντως ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ορθολογικοί. Και εδώ τίθεται το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων. Διότι υπάρχουν ε, κάποιοι αντικαθεστοτικοί που τάσσονται υπέρ της Δύσης και στους οποίους θα πρέπει να δείξουμε την ε, υποστήριξη ε, της Δύσης. Ασκούνται πιέσεις κατά την επιβολή του νόμου. Αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε αυτή η πολιτική δίωξη να πάρει τέρμα, να πάρει τέλος και πρέπει εμείς να δείξουμε προσήλωση και αποφασιστικότητα προς το στόχο αυτό. Σε άλλα θέματα και συμφωνώ με το είπε η κυρία Χάρμς, πιστεύω δηλαδή ότι εν γέννη μπορεί να έχουμε διαφορετικές θέσεις, τα κρατη δηλαδή, να έχουν διαφορετικές θέσεις, αλλά δεν πρέπει να επιβάλλουμε τις την πολιτική για τη σχέση μεταξύ των φίλων στις χώρες της γειτονίας. Της γειτονίας. Γιατί αυτό ισοδυναμεί με την υποστήριξη της πολιτικής του Πούτιν. Γιατί η Ρωσία εκμεταλλεύεται τη δική μας ιδεολογικά εμπνευσμένη υποστήριξη για να αποθαρρύνει τις χώρες αυτές από μια προσέγγιση προς τη Δυτική Ευρώπη. Απευθύνω λοιπόν έκκληση να είμαστε όσο δυνατόν πιο μέτριοπαθείς. Η πολιτική κρατούμενη βεβαίως είναι ένα θέμα καυτό. Πρέπει να απαιτήσουμε την αποφυλάκησή τους. Κύριος Παντσέρη, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κανιέτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος την μέσω του κυρίου Πρέντα και να σταθώ στην απόφαση του δικαστηρίου των, του Στρασβούργου για τον τέος Πρωθυπουργό. Η απόφαση αυτή επιδεικνύει ακόμα, απόδεικνύει για μια ακόμη φορά τον τρόπο που η πολιτική εξουσία ελέγχει τη δικαστική στη Γεωργία πολιτικά κίνητρα οδήγησαν στην κράτηση πριν από τη διεξαγωγή της δίκης, παραβιάστηκε το άρθρο 18 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι ήδη από πέρυσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε μία απόφαση για την περίπτωση του τέος Πρωθυπουργού. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής, σημειώνεται ότι σε διάφορα σημεία παραβιάστηκε η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και η απόφαση αυτή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να μας ανοίξει τα μάτια και να πιέσει την κυβέρνηση να πει ότι όχι μόνο να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να περιορίζεται στα λόγια συμμόρφωσης αλλά και στις πράξεις συμμόρφωσης. Η περίπτωση Μεραμπισβήλη είναι κάτι το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις αρχές της Γεωργίας και είναι δύσκολο να δεχθούμε την απόφαση ε, της, του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι η απόφαση αυτή θα οδηγήσει στην πληρωμή αποζημίωσης στον Μεραμπισβίλη, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι τέτοιου είδους δηλώσεις από πλευράς των εκπροσώπων της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Πρέπει να σταματήσει κάθε δίωξη εις βάρος του Μπεραβεσβήλη, θα πρέπει να απολυθεί αμέσως χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. από τη Διεύθυνση Γειτονίας και Μακροοικονομικής Βοήθειας. Thank you very much, uh, Chair. My name is Jan from the... Uh, Λέγομαι Ρίζα. από το τμήμα που ασχολείται με την οικονομική συνδρομή προς τις χώρες γειτονίας. Να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη για την υποστήριξή τους στη συγκεκριμένη μακροοικονομική βοήθεια προς τη Γεωργία. Η Γεωργία έχει επίγουσες ανάγκες για τα επόμενα τρία χρόνια και στα πλαίσια του προγράμματος του Δέλτα Νιτάφ. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται βασικά με τρεις παραγόντες, έλλειμμα τρεχουσών πληρωμών, εξωτερικό χρέος, ανάγκη αύξησης του αποθεματικού, του συναλλαγματικού και αύξηση των απαιτήσεων απόσβεσης ε, του χρέους τα επόμενα τρία χρόνια. Όλα αυτά τα θέματα μεταξύ τους βέβαια συνδέονται και όλα μαζί αποτελούν τη βάση της πρότασή μας για την βοήθεια προς τη χώρα αυτή. Τα 42 εκατομμύρια καλύπτουν το 1 τρίτο περίπου του κενού χρηματοδότησης προς τη Γεωργία και ότι δεν καλύπτεται δηλαδή από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Δέλτα Νιτάφ. Είναι μια καλή ισορροπημένη παρέμβαση διασφαλίζοντας αν θέλετε και τα συμφέροντα της Ένωσης και μοιράζοντας το βάρος μαζί με τους άλλους πιστωτές. Να επιστήσω την προσοχή σας και στην ανάγκη η απόφαση αυτή να ληφθεί παρακαλώ γρήγορα γιατί είναι ένα μέσο επαναλαμβάνω κατεπήγον και έχει ήδη υπάρξει αναφορά στο ελεγκτικό συνέδριο και στην απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναζητήσει ε, τρόπους συνεργασία με τους συνομοθέτες για να καλυφθούν οι απαιτήσει αυτές. Και ο Επίτροπός μας, ο κύριος Μοσκοβισή, αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης της συμφωνίας αυτής στα πλαίσια της ΣΥΝΤΑ πριν δύο εβδομάδες. Να αναφερθώ τώρα σε κάποια από τα θέματα που εσείς θέσατε λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά την προτινόμενη κοινή δήλωση Ταυτόχρονα να υπογραμμίσω πως εμείς από πλευράς της Επιτροπής δεν είμαστε ε, απόλυτα γνώστες του τι σκοπεύετε να πετύχετε μέσω της δήλωσης αυτής. Προφανώς δημοκρατία, κράτος δικαίου, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι και αλλιώς, ανήκουν σε κάθε νέα απόφαση. Αυτά τα υπενθυμίζει η δήλωση η αρχική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πέραν αυτού όχι. Κάτι το νέο. Από ό,τι φαίνεται πάντως, υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες οι οποίες έχουν τεθεί και για τη Γεωργία οι ανησυχίες αυτές δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό και εδώ με ελέγχει και η, ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πάντως νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι δύσκολα θα παρακρατούσε μια πληρωμή ε, προς τη Γεωργία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν έχει εκπληρώσει κάποιες προϋποθέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοιου είδους ε, οι επαναλαμβανόμενες καταθέσεις δηλώσεων ε, συνοδευτικά με ε, τα υπόλοιπα επίσημα κείμενα δεν είναι κάτι το υποχρεωτικά χρήσιμο. Βέβαια στην περίπτωση της Μολδαβίας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια ειδική περίπτωση αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας αν μια τέτοια δήλωση για τη γεωργία είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να υποτιμήσει αν θέλετε τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες δηλώσεις τις οποίες έχετε καταφέσει στην περίπτωση της Μολδαβίας. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι χρειάζεται μια τέτοια κοινή δήλωση. Τώρα για τα υπόλοιπα θέματα τα σχετικά με τις πολιτικές προϋποθέσεις και τα λοιπά σε σχέση με το άρθρο 2. Έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη εντολή για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις πολιτικές και τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Και το θέμα τώρα των πληρωμών και εδώ απαιτείται να υπάρξει μια πρώτη αξιολόγηση. Έχουμε λοιπόν από τη μία τις πολιτικές προϋποθέσεις, οι οποίες από για την απέτηση ενός τρέχοντος προγράμματος του ΔΝΤ είναι ε, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας. Από την άλλη έχουμε και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας. Να θυμίσω ότι το MFA είναι φυσικά ένα μακροοικονομικό μέσο συνδρομής και στόχος του είναι ακριβώς να μειώσει τα ευάλωτα χαρακτηριστικά και να αποφευθούν οικονομικές κρίσεις στο μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι όροι αυτοί συνδέονται και με το στόχους που έχει το συγκεκριμένο μέσο. Ε, παραπέμπουν επίσης και στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, του 2013 στο 1α για το μακροοικονομικά μέσα, εφαρμογή δηλαδή πολιτικών προγραμμάτων με ισχυρές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Αυτά όλα περιλαμβάνονται και στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 22 και στα άρθρα 3 που αναφέρεται στις οικονομικές, στην οικονομική συγκυρία. Η ισχύ λοιπόν και η δυνατότητα μόχλευσης του MFA ε, συνδέεται άμεσα με τον αρχικό στόχο του και γι' αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα σίγουρος, ε, επαναλαμβάνει ο ομιλητής, ε, να επιβαρύνουμε, υπέρ του να επιβαρύνουμε την αιρεσιμότητα με νέους τομείς και νέα θέματα. Οφείλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για μας, είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλά από τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σε συμφωνία αυτή συνδέονται άμεσα με τις οικονομικές εξελίξεις και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Βέβαια η Συμφωνία Σύνδεσης έχει ένα ορίζοντα εφαρμογής πολυετή, ενώ ε, το MFA είναι ε, κάτι το οποίο λειτουργεί υποχρεωτικά πιο βραχυπρόθεσμα και έχει σαν άμεσο στόχο να καταστήσει τις προϋποθέσεις ε, για περαιτέρω ανάπτυξη εφικτές. Αυτά. Ίσως να πω κάτι άλλο για την κατανομή ανάμεσα σε δάνεια από τη μία και ε, μη επιστρεφόμενες ενισχύσεις από την άλλη. Αυτά όλα εξαρτώνται και από το κατακεφαλήν εισόδημα της κάθε χώρας, όπως ακόμα και για τις δυνατότητες επιστροφής του χρέους. Η Γεωργία έχει κάνει πρόοδο σε σχέση με τους λογαριασμούς κατακεφαλήν εισοδήματος, σε σχέση με τα τελευταία προηγούμενα 5-10 χρόνια και γι' αυτό τα μη επιστρεφόμενα χρηματοδοτικά μέσα έχουν μειωθεί σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αντίστοιχες παρεμβάσεις μας οικονομικές. Αυτά. Και τώρα Πιο σύντομα μόνο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσθέσω να είμαι ο το πιο σύντομο. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι η Γεωργία είναι η χώρα της Ανατολικής Εταιρική Σχέσης που πλησιάζει περισσότερο αυτό που είχαμε κατά νου όταν ε, συστήσαμε ακριβώς ε, την Ανατολική Εταιρική Σχέση του 2008-2009. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και στην τελειότητα πολλά ε, θέματα που φτύξατε σήμερα μας βρίσκουν σύμφωνους. Υπάρχει και η έκθεση της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης που δημοσιεύθηκε μάλλον τον Νοέμβριο. Έχουμε και άλλους ε, στόχου του οποίους θα συζητήσουμε στι αρχέ του 2018 στο Συμβούλιο που εξετάζει ακριβώ την ε, Συμφωνία Σύνθεσης. Αναγνωρίζουμε και τη σταθερότητα και την αφοσίωση και προσήλωση της Γεωργία. Υπήρξαν εκλογέ στι 21 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου, τοπικές εκλογέ Και εν γέννη θεωρείται ότι ε, έγιναν σεβαστές οι διαδικασίες και η προλογική εξαρτία και οι πολιτικές ελευθερίες. Υπήρξαν διάφορες μεταρρυθμίσεις 2017, έχουμε πλέον και ε, καθεστώς απαλλαγής από ε, υποχρέωση θεωρήσεων από το Μάρτιο 2017. Σε ό,τι φορά τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση, χαιρετίζουμε τη, το, τις πρόσφατες τροπολογίες που συνάδουν πλήρω με τις συστάσεις της Επιτροπής Βενετίας. Παρακολουθούμε το συνέγγι και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού ε, τομέα καθώς και την ε, υπεράσπιση των ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων. Έχουμε και το συνήγορο του πολίτη που έκανε ένα γύρο διαβούλευσης γενικά με πολλούς εμπλεκομένους και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερότητα ε, των μεταρρυθμίσεων, γι' αυτό και είμαστε και υπέρ τη επιχείρηση αυτή. Εμεί, ω Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τι υπηρεσίε τη Επιτροπή και έχουμε αναφέρει ότι η αξιολόγησή μας παραμένει ενισχύ και ότι ε, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επιβεβαιώνουμε όμως εκ νέου ότι η υπηρεσία μας είναι τεθειμένη να παράσχει ε, λεπτομεριακή αξιολόγηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, καθόλου τον κύκλο του εγχειρήματο ε, τη μακροοικονομική συνδρομή. Έχουμε όμω κάποιε επιφυλάξει κατά πόσο είναι πραγματικά απαραίτητη αυτή η κοινή δήλωση, δεδομένου ότι η κατάσταση δεν είναι αντίστοιχη με αυτή στη Μολδαβία, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο δραματικά και όπου οι συστάσει δηλαδή τη Επιτροπή Βενετία δεν ε, έχουν γίνει σεβαστέ και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουν σεβαστέ και στο μέλλον. Οπότε σας καλώ να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ. Μαμίνκης. Ε, Ο εισηγητής. Thank you, Chair. Sorry, sorry. Metti le cuffie, se no non mi ascolti. Βάλε τα ακουστικά σου, όλες να μ' ακούς. Ο κύριος Γκρένς, ουσιαστικά, είπε ότι δεν έχει καταλάβει τι δουλειά κάνει Αν του το εξηγήσεις, να τον ικανοποιήσουμε κιόλας. Για άλλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω είπα, έχουμε στείλει πολλέ ερωτήσεις, έχουμε λάβει πολλές απαντήσεις, οι οποίε μας ικανοποιούν πλήρω. Τις έχουν λάβει τις απαντήσεις όλοι οι σκιώδεις και είπα ότι έχω καταθέσει μόνο μία τροπολογία. Δεν κατανοώ λοιπόν ε, περί τίνος πρόκειται. Με... Σαφέστατη η απάντηση και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι για τις τροπολογίες σας έχετε προθεσμία τις 7 Δεκεμβρίου και στις 23 Ιανουαρίου θα δούμε το θέμα στην Επιτροπή μας και έτσι τελειώνουμε το θέμα αυτό για απόψε. Λοιπόν, τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την απαλλαγή του Γενικού Προϋπολογισμού 2016 με εισηγητή τον Κριστιαν Πρέντα και του δίνω το λόγο. Από ό,τι βλέπω επικρατεί ταραχή στους ε, πρασίνους. Πάολο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι έχουμε ακόμα 13 λεπτά για τρία σημεία. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εξετάσω από κοινού τα ζητήματα της απαλλαγής. Ξεκινώ από την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017, 2016, νόμι για το τμήμα που μας ε, ε που μας αφορά εμάς, που είναι ο τομέας 4, έχουμε ε, σημαντική μείωση του ουσιαστικού σφάλματος σχέση με το 2015, 2,8%, πήγαμε στο 2,1%. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη και ελπίζω και στα επόμενα χρόνια να πέσουμε κάτω από το 2% και συνιστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει όλες τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου γιατί ε, φάνηκε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πτώση του 0,7% εάν είχαν αξιοποιηθεί ε, γέρος όλες αυτές οι πληροφορίες. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τις ε, αποστολές που έγιναν στο πλαίσιο της ε, κοινή πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας και χαιρετίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτάχυνση των προσπαθειών τη. Υπάρχει ένα τελευταίο σχέδιο σε ό,τι αφορά την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τις αδυναμίες στις ελεγκτικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες χώρες που είναι υποψήφιες ή ενδεχομένως να γίνουν υποψήφιες και επειδή δεν υπάρχουν αυτές μάλλον οι υγροτικές αδυναμίες κατόπιν σύσταση και του ελεγκτικού συνεδρίου, νομίζω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να επιμείνει στην βελτίωση ε, της διαχείρισης αυτών των λογιστικών ελέγχων. Γι' αυτό προτείνω αλλαγή στην παράγραφο 4 που θίγει αυτό το σημείο. Νομίζω ότι χρειάζεται ε, σαφέστερη διατύπωση ότι αφορά την αιτία του προβλήματος που είναι ανεπάρκεια της λειτουργίες στα ελεγκτικά συστήματα κάποιων από τους εταίρους μας. Για τα υπόλοιπα σημεία, το σημείο 5 για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, με τα χαράς βλέπω ότι ο διοικητικός προπολογισμός αυτού του θεσμικού οργάνου εκτελέστηκε χωρίς ε, ε, σημαντικό ουσιαστικό σφάλμα. Ε, ωστόσο, ευχαριστώ την προσοχή σας στο γεγονός. Τι έγινε ξαφνικά, φύγαν όλοι. Με το που φτάνουμε στον προπολογισμό, βλέπω ότι μόνο εγώ μένω. Και εσείς κύριε Πρόεδρε βεβαίως. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ε, ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους για να ε, αντισταθμίσουμε τις υφιστάμενες λειτουργίες σε ό,τι αφορά ε, τους ανθρώπινους πόρους, τα νέα ή και παλιότερα κράτη-μέλη και την καλύτερη λειτουργία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα, τα αναπτύξω και στην έκθεση που θα σας υποβάλω. Ε, θέλω να πιστεύω την προσοχή στο γεγονό ότι το νομικό συνέδριο έχει εντοπίσει ανεπάρκειε και αδυναμίε ε, ό,τι αφορά τι ε, δημόσιε συμβάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πρόκειται για κάτω από 70.000 ευρώ. Και προτείνω να υιοθετηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αφόσον έθιξε το ζήτημα των ανθρωπίνων πόρων, θα ήθελα επίση να σταθώ στη σημασία του καλύτερου προσδιορισμού του περιεχομένου των νέων πολιτικών και λέω ότι πρέπει να συνοδεύονται και με δημοσιονομικούς πόρους που θα επιτρέψουν στα θεσμικά μας όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης, να τα υλοποιήσουν. Εδώ βέβαια πρόκειται για ένα ε, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να θίξουμε κυρίως στο πλαίσιο της ε, κατάρτισης του σχεδίου προπολογισμού και του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω και εδώ. Αυτά σε αδρές γραμμές για τις δικές μου ε, εκθέσεις. Ε, μέχρι 7 Δεκεμβρίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίε και βεβαίω ε, θα συνομιλήσω και θα συνεργαστώ με τους σκιώδει εισηγητές που ελπίζω κάποια στιγμή τουλάχιστον να εμφανιστούν και στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ ο όρο σκιώδη ε, παίρνει όλη του την ε, κυριολεκτική σημασία. Είναι πραγματικά σκιώδη οι απόντε συνάδελφοι. Για να δούμε η κυρία Νικόλ Σμιτ από την Κομισιόν, παρακαλώ. Νικόλ Σμιτ... Ε, υπεύθυνη με το, για τη σχέση με το Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και με τις ελεγκτικές αρχές ε, σε θέματα προπολογισμού από τη Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ για τα σημεία που αναφέρατε. Ιδιαίτερα θέλω να καλύψω το θέμα των ελεκτικών αρχών. Τα, οι στάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου ακολουθούν ε, τη δουλειά της, της μονάδας μου που εντοπίζει αδυναμίες σε σχέση και με τις υποψήφιες χώρες και βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην επαλήθευση των δαπανών, αλλά διαπιστώνουμε και βέβαια οι ελεκτικές αρχές ε, ότι υπάρχουν προβλήματα στις δομές και απουσία δεξιοτήτων, αλλά και οργανωτικού δυναμικού, προγραμματισμού, προσωπικού στις ελεγκτικές υπηρεσίες με τον οποίο τις επικεφαλής εγώ συναντήθηκα. Ακολουθούμε τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου ε, για να λύσουμε όλα τα ζητήματα, τα σχετικά με τις ελεγκτικές αρχές, αλλά παραμένουν προβλήματα σε σχέση με ορισμένε χώρες. Η κατάρτιση αλλά και οι προσλήψεις του ελεγκτικού προσωπικού συνεχίζονται, δίνουμε ε, κατευθυντήριες γραμμές, βελτιώνουμε τον προγραμματισμό και στη δική μου Γενική Διεύθυνση έχουμε ξεκινήσει μια επισκόπηση λεπτομερή των ελεκτικών αρχών στο σύνολό τους, με τις πληροφορίες που μας δώσαν αλλά και με μας ε, αυτοψίες προγραμματίζουμε, ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα δράσης για κάθε χώρα με βάση τις αδυναμίες και μια πολύ λεπτομερή επιτήρηση, αξιολόγηση κινδύνου, πρόγραμμα εργασίας των ελεκτικών αρχών. Και επίσης κάνουμε και workshop σε σχέση με τις διάφορες χώρες για να ανταλλάξουμε βέλτιστες ε, πρακτικές, όπως είχαμε παραδείγματα τη δυνατότητα με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πρόσφατα, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των διαφορών ελεκτικών αρχών και να ανταλλάξουν απόψη. Το ελεκτικό συνέδριο παρακολουθεί ε, βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα και ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο το περιθώριο του ποσοστό του σφάλματος, να βελτιωθεί το δυναμικό των αρχών. Βεβαίως και δεχόμαστε τις επικρίσεις και είμαστε σε, στη διάθεση του Κοινοβουλίου όπως και του Ελεκτικού Συνοδρίου για να βελτιώσουμε τις ελεκτικές μας δραστηριότητες. Ευχαριστώ τελεία. Να δώσω τώρα το λόγο. Υπεύθυνο τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ και η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ είναι ικανοποιημένη από την πτώση του ποσοστού των λαθών σε 2,1 από 2,8. Συνολικά το ποσοστό αυτό χαμηλώνει για πέμπτο συνεχές ε, ε, έτος πέρα από τους στόχους που είχαν τεθεί, όλοι αυτοί είναι καλοί δείκτες προόδου. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης. Εφαρμόζουμε τις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου στο σημείο 3 και μετά από αυτά που είπε ο εισηγητής. Ασχολούμεθα και με το θέμα των επιδοτήσεων. Έχουμε καταθέσει κάποιες επιφυλάξεις μας ε, για την ετήσια έκθεση σε σχέση με τα προγράμματα δράσης και την άμεση διαχείριση, όπως και την αναθεώρηση των όρων αναφοράς για τις ελεγκτικές διαδικασίες, την, τον έλεγχο και την εποπτεία και διάφορες δράσεις που αναλαμβάνουν οι διάφορες υπηρεσίες στον τομέα της κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχνεύουν τα σωστότα τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα λάθη. έτσι ώστε να καλυφθούν οι αδυναμίες τις οποίες έχει εντοπίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Και φυσικά και υπάρχουν πάντα και οι διαδικασίες ανάκτησης, οι οποίες ε, όταν χρειάζεται θα τίθενται σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ η κυρία Κάμπελ οριζόντια διαχείριση πολιτικών. Good afternoon, Mr. Chairman, and thank you for the opportunity to give a few brief remarks. I'm... Ευχαριστώ για στα πλαίσια της νέας αυτής υπηρεσίας, της εξωτερικής υπηρεσίας να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα σχόλιά του και για το επίπεδο λαθών στο οποίο υπήρξαν προσπάθειες σε σχέση με το ισοζύγιο του ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς είμαστε υπέρ της ισορροπίας σε επίπεδο φύλων, προέλευσης κτλ. Να πω ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας κ. Σμιτ έχει δημιουργήσει ένα task force για την ισότητα των ευκαιριών και ταυτόχρονα έχουμε και την πρώτη στρατηγική για την ισότητα ευκαιριών ανδρών γυναικών στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Για τα θέματα των προμηθειών θα εφαρμόσουμε τις αλλαγές από του χρόνου θα προχωρήσουμε και σε συμπληρωματικές μορφές κατάρτισης έτσι ώστε να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται. Είπατε λοιπόν κύριε Πρέντα ότι η 7η Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Κλείνουμε για λίγη ώρα και περιμένουμε για την επόμενη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, 7, σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη για σήμερα και καλωσορίζω τον Υπουργό Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας Αλβανίας, τον Ντίτμιρ Μπουσάτη, που όλοι βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά. Καταρχάς, σας συγχαίρουμε για την 105η επέτειο της ε, ανακήρυξης ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, κύριε Μπουσάτη, για αυτό το διάλογο. Μετά βέβαια την εισαγωγική σας παρέμβαση θα σας δώσω το λόγο για ερωτήσεις στους συναδέλφους. Ε, περιμένουμε τα σχόλιά σας για την ε, πολιτική κατάσταση τις ε, μεταρρυθμίσεις, ε, το ρόλο της δικαστικής εξουσίας και βέβαια την περιφερειακή συνεργασία με τους εταίρους σας. Έχει άνετη πλειοψηφία η κυβέρνησή σας και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τις ε, μεταρρυθμίσεις, αλλά πάλι έχει την αντιπολίτευση, τη δικαστική εξουσία αλλά και την κοινωνία των πολιτών που πρέπει να πείσει για την εξασφάλιση ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος. Περιμένει μάλιστα την απόφαση για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων ε, για την ημερομηνία εκείνης των, συνομιλιών για την προσχώρηση, ανεξάρτητος του εισέκβαση αυτής της απόφασης, πρέπει να συνεχιστούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, γιατί, κυρίως για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως ε, του προβλήματος των ναρκωτικών και βέβαια πρέπει να επενδύσετε οπωσδήποτε και σε καλές σχέσεις γειτονίας. Αυτά από πλευράς μου και περιμένω τις δικές σας θέσεις κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μαζί σας σήμερα. Γνωρίζω ότι είμαι στον σωστό χώρο για να αναφερθώ στο θέμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο ρόλος των κοινοβουλευτικών και ιδιαίτερα της Επιτροπής σας είναι καθοριστικός για την θεσμική και δημόσια στήριξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, η επικοινωνία και η διαφθρωτική συνεργασία μεταξύ μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στο κλίμα σκεπτικισμού που επικρατεί γύρω από τα θέματα των διευρύνσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις επιρροές που μπορεί να έχει σε μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε τη μοίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η δική μας μοίρα φυσικά εξαρτάται από τις δικές σας προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη Ευρώπη. Γνωρίζετε ότι οι λαοί των Δυτικών Βαλκανίων εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν επενδύσει σε ένα όνειρο το οποίο τώρα έχει γίνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σύνδεσης και ένωσης με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν επιθυμούμε πλέον νέες διαχωριστικές γραμμές. ανεξαρτήτως ε, του εισοδήματός τους ή των ιδεολογιών τους, οι κάτοικοι της Αλβανίας συνδέουν την Ευρώπη με την ειρήνη, την ανάπτυξη και την ευημερία. Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει βιώσει 15 χρόνια χωρίς καμία βίαιη σύγκρουση, υπάρχει πολιτική ορίμανση, σχέσεις με τα κράτη-μέλη και η δυναμική των νέων προσπαθειών ολοκλήρωσης της συνεργασίας έχει βοηθήσει σταδιακά στο να δινήξουν νέες προϋποθέσεις για τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες της περιοχής. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε βοηθήσει επίσης και την απόκτηση αίσθησης ιδιοκτησίας των προσπαθειών συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Γι' αυτό λοιπόν συμμετέχουμε σε κοινά προγράμματα και βλέπουμε το μέλλον μας όχι σαν μια δυνατότητα να κερδίσουμε κάποιο παιχνίδι εις βάρος του άλλου, αλλά να μοιράσουμε όλοι τα κέρδη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προοπτική ένταξης είναι βασική ε, στόχευση της κυβέρνησης μας, κάτι το οποίο έχει σαν στόχο να κρατήσει την περιοχή μας ειρηνική και σε στενή συνεργασία τα επίπεδα συνεργασίας ανάμεσά μας ε, ε, έχουν αποδείξει τα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Ε, η συμπερίληψη λοιπόν της Αλβανίας γεωστρατηγικά είναι βασικός στόχος για τις υποψήφιες χώρες. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι η σωστή επιλογή και είναι μια επιλογή χωρίς καμία εναλλακτική. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι καθυστερεί και γι' αυτό μπορεί να ε, γίνει κάτι το απρόβλεπτο στο μέλλον. Μπορεί να καταλήξει σε μια τεχνική διαδικασία χωρίς τέλος, χωρίς ε, μια ημερομηνία, χωρίς ένα χρονικό όριο. Κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες, δυσφορία στους νέους κυρίως και τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας μου. Υπάρχουν επίσης και διάφορα περιφερειακά θέματα με δυνητικά αποσταθεροποιητικές συνέπειες. Και γι' αυτό λοιπόν το πολιτικό βάρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης είναι καθοριστικό. Το να σκέφτεται κανείς τα θέματα αυτά στρατηγικά σημαίνει ε, να υπολογίσει το κόστος της μη ένταξης, ιδιαίτερα όταν το συγκρίνει με το μικρό κόστος της ένταξης των χωρών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικά σε σχέση με την διεύρυνση, λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία τρίτων παικτών στα Δυτικά Βαλκάνια και κάποιων σιωπηλών στην φάση αυτή εξωτερικών απειλών. Τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να ειδωθούν όχι σαν μια διεύρυνση της Ευρώπης, αλλά σαν ένας καθοριστικός παράγων ασφαλείας. Αυτό που κάνουμε και σαν μέλη του ΝΑΤΟ συμβαδίζει με αυτό τον στρατηγικό τρόπο σκέψης. Και νομίζω ότι η συνεισφορά μας ως υποψηφίας χώρας θα είναι σημαντική στο νέο πλαίσιο ασφαλείας της Ευρώπης. Αυτά έχουν σημειωθεί και από τους εκπροσώπους της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον πρόεδρο Ιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης για μια αξιόπιστη προοπτική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και για μια νέα πρόταση για την περιοχή αυτή τον μήνα Φεβρουάριο. Σημειώνουμε με ικανοποίηση και τα στοιχεία του Πρόεδρου Μακρόν στο ετήσιο μανιφέστο του ότι τα Βαλκάνια θα είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμούμε ιδιαίτερως και τις δηλώσεις της κυρίας Μογκερίνη. Τέλος, εκτιμούμε επίσης και τις βασικές για μας θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας. Όμως όλα αυτά δεν αρκούν. Το όραμα της ένταξης και της στρατηγικής σημασίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, η διεύρυνση θα πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει στην ατζέντα των κοινοτικών υποθέσεων. Περιμένουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη για το πώς θα καταλήξουμε στην έναρξη των διαπραγματεύσεων. Πώς θα δώσουμε διαφάνεια και αξιοπιστία, πώς θα προσδώσουμε διαφάνεια και αξιοπιστία. Η Αλβανία είναι υποψηφία χώρα από το 2014 και μια τέτοια απόφαση έναρξης των διαπραγματεύσεων θα είναι μια ιστορική στιγμή για τη μορφοποίηση και τον εξυγχρονισμό του δημόσιου μηχανισμού θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τους διοικητικούς ε, τρόπους λειτουργίας της χώρας και θα βοηθήσει επίσης και τη σωστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των, της δικαστικής εξουσίας. Η κυβέρνηση της Αλβανίας λοιπόν θα συνεχίσει την μεταρρυθμιστική της ατζέντα, ιδιαίτερα στον τομέα του κράτους δικαίου. Είναι βασικός πυλώνας ε, εγκαθίδρυσης μιας δημοκρατικής κοινωνίας, μιας λειτουργούσης ε, οικονομίας. Εμείς ε, και η μεταρρύθμιση, την οποία, μάλλον η μεταρρύθμιση την οποία εμείς εφαρμόζουμε στον τομέα της δικαιοσύνης είναι καθοριστική και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από διεθνή εποπτεία. Τα αποτελέσματα εις βάρος του διεθνούς εγκλήματος και λαθρεμπορίου ε, κάναβης ε, είναι βασικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε πετύχει. Η συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές της χώρας και ε, στις αστυνομικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω πορεία ολοκλήρωσης και ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα κεφάλαια 23 και 24. Ο βελτιωμένος πολιτικός διάλογος μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε σε βασικές αλλαγές και στο συνταγματικό χάρτη της χώρας, και να πάρουμε εν πάση περιπτώσει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης τον Ιούνιο του 2017 η σωστή διεξαγωγή των εκλογών, όπως επίσης και η υιοθέτηση τριών βασικών νόμων με διακομματική στήριξη σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για την επαναξιολόγηση των, των δικαστών δεν θα ήταν κάτι το θετικό χωρίς ε, την ύπαρξη αυτού του βελτιωμένου πολιτικού διαλόγου. Να πω ότι η Αλβανία ήταν σαφής σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε στις ίδιες αξίες. Σαν σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Αλβανία δεν θεωρεί ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Η Αλβανία είναι, συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου κατά 100%. Η Αλβανία είναι υπερήφανη επίσης γιατί ήταν μια από τις πρώτες χώρες που αντέδρασε στις κινήσεις του ΝΤΑΕΣ στην περιοχή και των ακραίων εξτρεμιστών. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την περιφερειακή συνεργασία. Είναι, έχουμε τα μέσα για να μετατρέψουμε την περιοχή σε μια πραγματική δημοκρατική ζώσα και περιοχή. Ε, επίσης έχουμε και πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης της οικονομικής συνεργασίας μετά από τη συνάντηση κορυφής το καλοκαίρι του 17 στο διράχιο Να κλείσω λέγοντας το ότι ε, η περιοχή αυτή περιβάλλεται από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν ανήκει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ε, δίνει δυνατότητες κίνησης σε τρίτους και πολλές φορές υπάρχουν προπαγανδιστικές ε, ενέργειες από διάφορες χώρες στην περιοχή. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν πρέπει να παρεμποδίσει την ένταξη της περιοχής στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία σαν παράδειγμα δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή αλλά και δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Παρ' όλα αυτά έχει την δυνατότητα να παρεμποδίσει τις διαδικασίες. Η περιοχή μας όμως χαρακτηρίζεται από περιπλοκότητες. Κάποιες, μέλη είναι, κάποιες χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, κάποιες άλλες θέλουν να γίνουν γρήγορα, κάποιες είναι σε ε, επίπεδο διαπραγμάτευσης, δύο είναι υποψήφιες, δύο στοκεύουν στο να γίνουν υποψήφιες, παράλληλα και με απειλές οι οποίες προέρχονται από κάποιες από τις χώρες αυτές καθιστούν την περιοχή και την Αλβανία καθοριστικές για την γεωπολιτική ισορροπία της Ευρώπης και της διατλαντικής συνεργασίας. Η επιτάχυνση λοιπόν των διαπραγματευτικών διαδικασιών θα αποδείξει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με αποτελεσματικότητα σε λειτουργικές μορφές συνεργασίας. Η Αλβανία έχει ανάγκη και της αξίζει να περάσει στην επόμενη φάση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε από τους εταίρους μας να κάνουν και αυτοί ό,τι απαιτείται. Ελπίζουμε ότι το 2018 θα είναι αποφασιστικό έτος για την Αλβανία. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα δείξει τις σωστές κατευθύνσεις για και θα επιβεβαιωθεί και θα επιβαβευθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια την οποία κάναμε μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν απαραίτητο το 2018 μαζί με τη δική σας βοήθεια μια αποφασιστική χρονιά για την Αλβανία. Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παραμείνει η κινητήρια δύναμη για την πρόοδο και το μέλλον της περιοχής μας. Thank you, Ευχαριστούμε τον κύριο για τα όσα μας είπε για την κατάσταση στη χώρα του, ιδίως ό,τι αφορά την διαδικασία της διεύρυνσης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Φλέκενστάιν, παρακαλώ. Ε, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την ομιλία του. Θα ήθελα να συνεχίσω στα γερμανικά, Äh, Entschuldigung. So, äh, ich Λοιπόν, σε πολλά σημεία, κύριε Υπουργέ. Έχετε πολύ εύστοχα επισημάνει ότι πρέπει να υλοποιηθεί το όραμα και θα προσθέσω και το αντίστροφο ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να κάνετε εσείς καλά τη δουλειά σας στη χώρα σας αυτές με αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα γειτονικά σας κράτη για τα οποία γίνεται λόγος για διαδικασία ένταξης να αποδειχθούν αξιόπιστη εταίρη. Αξιόπιστος εταίρος σημαίνει προσδορίζω προϋποθέσεις, εάν δεν πληρούνται δεν μπορείτε να περιμένετε τίποτα, εάν πληρωθούν όμως τότε πολύ σωστά θα πρέπει να έχετε και εσείς την προσδοκία ότι θα δείτε την ανταμοιβή και γι' αυτό θεωρώ όπως και εσείς ότι το 2018 πρέπει να ξεκινήσουν πρέπει να ξεκινήσουν, υπογραμμίζω πρέπει να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με την Αλβανία, όχι γιατί θα έχουν ρυθμιστεί τα πάντα και θα κλείσει έτσι πανηγυρικά ε, η διαπραγμάτευση, αλλά γιατί θέλουμε επιτέλους να δούμε την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης και γιατί η κυβέρνηση αλλά και του Κοινοβούλου συμπεριλαμβανομένης και της ε, αντιπολίτευσης έχουν κερδίσει αυτό το βήμα και με τη μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας που έχει έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες η Αλβανία, αλλά και γιατί οι προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχουν μπει σε σωστό δρόμο. Για το οργανωμένο έγκλημα ξέρουμε ότι μένουν ακόμα αρκετά να γίνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επισημάνει πολλά ζητήματα στην κυβέρνησή σας. Έχουμε και στις δικές μας χώρες εγκληματικότητα, η οποία όμως πολλές φορές έχει τις ρίζες της στην Αλβανία. Και υπουργοί από διάφορες χώρες, κατοχώρες, Γερμανία, επεξεργάζονται το πρόβλημα αυτό. Βλέπουμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουν να βλέπουμε καλά αποτελέσματα. Και γι' αυτό, για να ολοκληρώσω με πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση, ε, γιατί πολύ συχνά λαμβάνω επιστολές, ε, τηλεφωνικά μηνύματα, όπου κάποιος πολίτης μου καταγγέλει κάποιο πολιτικό ή κάποιος από την αντιπολίτευση. Οι παραδείγματοι μου αναφέρουν τον Υπουργό των Εξωτερικών όχι μόνο ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο εισαγγελέα από το Κοινοβούλιο ή και άλλη περίπτωση με τον εισαγγελέα όπου πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μπαίνουν από λογαριασμού του εξωτερικού στη χώρα για να χρηματοδοτήσουν την προεκλογική εκστρατεία. Ε, δεν είναι τόσο ότι πιστεύουμε τις καταγγελίες ως έχουν, αλλά μας ενδιαφέρει να μπορεί η εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Και εδώ ακριβώς βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Μια τελευταία κουβέντα. Η δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο και η Κυβέρνηση και δεν το λέω ως Γερμανός βουλευτής όχι ο συγητής. Σημαίνει ότι πρέπει και να δοθεί η εκκίνηση για τις συνομιλίες του 2018. Κάθε άλλη απόφαση θα ήταν μεγάλο λάθος. Ευχαριστώ τον κύριο Φλέκινστάιν. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό ε, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας για αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αλβανία στην ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόκειται για διαφεσβήτητη πρόοδο και αναμφίβολα όπως και τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια και η Αλβανία θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, να ε, προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Προσωπικά, μάλιστα, θεωρώ ότι και από δική μας πλευρά θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να θέσουμε μία προθεσμία. Προς το παρόν βρισκόμαστε στη φιλοσοφία του εντάξει κάποια στιγμή μακάρι να. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να θέσουμε ε, το 2025 ως προθεσμία για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά αυτό είναι δική μου προσωπική γνώμη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα της επικαιρότητα. Τι γίνεται με την διαδικασία που αφορά τους δικαστές. Ξέρω ότι υπάρχει, τρέχει μάλλον η πρώτη φάση, πότε θεωρείται ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί αυτό συνδέεται βέβαια και με το νέο γύρο διαπραγματεύσεων Δεύτερον, επειδή εγώ συμμετείχα σε αυτή την ε, αποστολή εκλογικών παρατηρητών που επί επιτόπου ε, παρακολούθησε τις ε, τελευταίες εκλογές, θα ήθελα να πείτε τι γίνεται με τις συστάσεις που έκανε η Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά και τον αρμόδιο οργανισμό και κατά πόσο υπάρχουν εξελίξεις. Και τέλος, για την κάναβη. Γιατί τελευταία έχουμε δει όλη αυτή και πάλι τη συζήτηση για την κάναβη μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας. Τι έχετε να μας ανακοινώσετε ως θετικό, θετική εξέλιξη για ένα φάκελο που πραγματικά είναι ιδιαίτερη σημασία για πολλούς Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κρίστιαν. Επόμενος ομιλητή Μπάστιαν Μπέλντερ για το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Γιατί είμαι και εισηγητής για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η Σύνοδος ε, στην Βουδαπέστη. Η Αλβανία ε, συμμετέχει σε αυτή τη μορφή συνεργασία μεταξύ ε, χωρών δυτική και ανατολική και Κεντρικής Ευρώπης και Κίνας. Ποιος είναι ο σκοπός, ποιοι είναι οι στόχοι της Αλβανίας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Κίνα. Με προσοχή ακούσαμε αυτά που είπατε, ότι ε, είστε υπέρ της ενότητας στην Ευρώπη, όμως ο τύπος ε, αναφέρει ότι εδώ στο Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου από πλευράς σοσιαλιστών, καθώς και πρόεδρος του ΕΛΚ, έχουν κάποιους, κάποιες επιφυλάξεις. Οπότε, ποιοι είναι οι στόχοι της ε, Αλβανίας και αφορά τις στενές της σχέσεις με την Κίνα και επίσης μήπως δημιουργείται εντάσεις σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή σας ένταξη δεδομένου ότι ε, ακολουθείτε πλήρως ε, την Κίνα και τις προοπτικές της, γιατί εμείς ε, εδώ εξετάζουμε κατά πόσο υπονομεύεται η συνοχή της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί εμείς είμαστε αλληλεγγύα, αλλά πρέπει να είστε και εσείς. Και δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι ασχολούνται μόνο με την Αλβανία και με τα συμφέροντά τη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέλτερ. Τώρα από πλευρά Πρασίνων, ο κύριο Πεσόλτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσίαση. για έναν ποταμό στην Αλβανία που είναι από τους μεγαλύτερους, 245 χιλιόμετρα συνολικό μήκος, έναν από τους τελευταίους μεγάλους ε, πραγματικούς ποταμούς ε, στην Ευρώπη. Η αλβανική κυβέρνηση έχει ε, παραχωρήσει τα δικαιώματα κατασκευής ε, μεγάλων έργων στον ποταμό σε αντίθεση με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αντίθεση και με αιτήματα των κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Το Κοινοβούλιο ανέφερε αυτό το ζήτημα και στο ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου του 2017 και αναδεικνύεται εκεί αυτό το ζήτημα και απευθύνεται και έκκληση προς την κυβέρνησή σας να επανεξετάσει ε, τη θέσπιση αυτού του εθνικού πάρκου ε, σε όλο το μήκος ε, του ποταμού και να εγκαταλείψει τα σχέδια για την κατασκευή νέων υδροελεκτρικών σταθμών στον ποταμό. Υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς αυτό για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες. Ένας ακόμη ομιλητής, ο κύριος Κουκάν. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι, ο κύριος Κουκάν τελευταίος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω κύριε Μπουσάτη. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η χώρα σας προοδεύει στον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η προσωπική μου εμπειρία λέγει ότι η χώρα σας αλλάζει, η Αλβανία αλλάζει, η Αλβανία επιτυγχάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα στην οδό της μεταρρύθμισης και έρχεται πιο κοντά στην ιδιότητα του υποψηφίου μέλους. Όπως είπε και ο κύριος Φλέκενστάιν, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Ξέρετε ε, ποιες είναι οι εκκρεμότητες από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις εκκρεμότητες αυτές οι κυβέρνηση σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα προχωρήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πρόσφατα τη στάση μας απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια, να είμαστε πιο υπεύθυνοι απέναντι στην περιοχή αυτή και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των συναδέλφων στις χώρες αυτές. Νομίζω ότι η περίπτωση της Αλβανίας θα μας το επιτρέψει να το αποδείξουμε αυτό. Ας ε, περιμένουμε λοιπόν θετικά αποτελέσματα και θετικές εξελίξεις για το 18 <clears throat> για την Αλβανία το θέμα είναι να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα στην διαδικασία γυτνίασης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω η χώρα να είναι έτοιμη για να το πετύχει αυτό και νομίζω ότι και εμείς σαν ΑΦΕΤ οφείλουμε να ρίξουμε το βάρος μας πίσω από τις συστάσεις τις οποίες θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα και να συνεργαστούμε σωστά με την χώρα σας. Ευχαριστώ κύριε Κουκάν. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από τους συναδέλφους. Να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Είχαμε αρκετές συζητήσεις στο παρελθόν για τη λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια και θα ήθελα και την άποψη της κυβέρνησης στα Τύρανα. Πώς βλέπετε εσείς τη διαδικασία του Βερολίνου, τι πηγαίνει καλά και τι μπορεί να βελτιωθεί. Και τι περιμένετε για την επόμενη συνάντηση στη Σόφια. θα ήθελα να πω ότι έχετε μέχρι 20 λεπτά για να απαντήσετε. Θα είμαι σύντομος και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, για τη διαδικασία μεταρρύθμισης που έχουμε ξεκινήσει στην Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ που διατηρείτε ζωντανή την ε, διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, όπως είπα και πριν, ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια, η περίπτωση της Αλβανίας είναι και ένα υπόδειγμα εκδημοκρατισμού και κίνητρο για μετάλλαξη. Θα δώσω απαντήσεις ε, σε έναν από τους συναδέλφους, τους βουλευτές, για τη δικασία επαλήθευσης ε, ε, για τους δικαστές και εισαγγελείς και των προκογών τους. Αυτό που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις μπορεί να ζούμε στα Βαλκάνια και η, Αλβανία να είναι τόσο μεσογειακή όσο και βαλκανική χώρα. με ως συνέπεια μια πολλωμένη πολιτική σκηνή και εσείς έχετε καταστεί μάρτυρας των προσπαθειών να, μας, να βρούμε μια βοήθεια για συμβασμό πριν τις εκλογές του Ιουνίου. Η πολιτική ε, αντίληψη έχει εμπλουτιστεί και το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει με την ψήφο του τη θέσπιση των σωμάτων επαλήθευσης και προαγωγών και άρα έχουμε δικαστές του Ανώτατου και του Σταγματικού Δικαστηρίου στις επιτροπές αυτές και εισαγγελείς του ψηλότερου επίπεδου, εισαγγελείς Αριού Πάγου του ΣΥΠΜΗΝ, και έχουμε τις πρώτες υποθέσεις ε, ε, ε μέχρι το, την άνοιξη δε πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια αξιόπιστη διαδικασία επαληθεύσεως από τις επιτροπές αυτές, τουλάχιστον για τους ε, ανώτατους δικαστές. Ε, σας ευχαριστώ πολύ όλους και τις κυβερνήσεις βεβαίως ε, που έχουν στηρίξει αυτή τη διαδικασία και τι βέβαια οι αποφάσεις που θα ληφθούν είναι αποφάσεις των ε, μελών των Επιτροπών, Αλβανών δηλαδή πολιτών, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχουν επωφεληθεί από την εμπειρία και τις γνώσεις ε, που τους προσφέρουν οι δικαστές ε, που έχουν επιλεγεί από δημοκρατικές διαδικασίες για σε σχέση με τις συστάσεις της, του ΩΣΑ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο εξελίξεις. Καταρχάς για την πολιτική βούληση για συνεργασία με τους ειδικού της ΟΝΤΙΡ και με τα διάφορα σώματα ώστε να βοηθηθούν οι διάφορες δομές να δώσουν απαντήσεις στα διάφορα θέματα και βέβαια η εγκαθίδρυση της ε, Επιτροπής Ad Hoc στο Κοινοβούλιο, διμερίους Επιτροπής, με συμπρόεδρο από την, συμπρόεδρους από την ε, συμπολίτευση και την αντιπολίτευση και πλαισιωμένους από ειδικού της ΟΝΤΙΡ. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι συστάσεις του ΩΣΑ και της ε, που έχουν να κάνουν με την αποπολιτικοποίηση της διαδικασίας που είναι κρίσιμοι τομής και απαιτούν όχι μόνο νομοθετική παρέμβαση αλλά και πολιτική βούληση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και περνώ στο τρίτο θέμα, καλλιέργεια κάναβης και ναρκωτικών. από την ε, πανηγυρική μας νίκη και ανάδειξη στην εξουσία. Αυτό ήταν ο αγώνα στον οποίο αποδεθήκαμε με την εντατικοποίηση του ε, αγώνα για την καταπολέμηση της κάναβης. Είπα και σε αγωγικές μου παρατηρήσει ότι ίσω είναι μοναδική περίπτωση η Αλβανία όπου σε συνεργασία με τους Ιταλούς της Guardia di Finanza έχουμε κάνει μαζικές επεμβάσεις και επιχειρήσεις και μπορούμε να μιλούμε πλέον για εκρίζωση των φυτιών κάναβης. Την δε στρατηγική και στόχευση της πρόληψης της καλλιέργειας της κάναβης τώρα μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε αγώνα κατά του εμπορίου, του λαθρεμπολιού της κάναβης. Βέβαια σας πενθυμίζω ότι είναι περιφερειακό το φαινόμενο, ένα φαινόμενο που άλλωστε δεν γνωρίζει σύνορα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, κυρίως τους ε, γειτονές μας που επηρεάζει το φαινόμενο και είμαστε βέβαια και στη διαδικασία της αντιμετώπισης των, της ρίζας του κακού, δηλαδή οικονομικές συνθήκες και γενικά ευημερία των πολιτών. Τέταρτη ερώτηση. Κίνα. Διμερείς σχέσεις. Ήταν σαφής νομίζω η τοποθέτησή μου πως η Αλβανία έχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποδείξει και επιδείξει στρατηγική σαφήνεια ως προς την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και δεν έχουμε την πολυτέλεια να στηριζόμαστε σε δύο καρέκλες όπως κάποιοι από τους γειτονέ μας. Σε αυτό είμαστε απόλυτα σαφείς. Από την άλλη, η παρουσία της Κίνας στην περιφέρεια ε, συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας δεν είναι για μας κίνδυνος, δεν είναι απειλή για την οικονομία μας, εφόσον και στο βαθμό που αυτή η οικονομική συνεργασία αναπτύσσεται με βάση τους κανόνες που έχουν οριστεί και επιβληθεί από το θεματολόγιο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η ευθογράμμιση της νομοθεσίας και των πολιτικών ακολουθεί ένα μόνο δρόμο, μία μόνο επιλογή, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ποταμός Ρώσα Πολύ σωστά είπατε ότι είναι μια συζήτηση που, μια απόφαση μάλλον που λήφθη κατόπιν ε, εντατικών συζητήσεων. Διάφορες ε, ομάδες πολιτών είχαν εκφράσει ανησυχίε για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα είναι υπό αναθεώρηση η απόφαση. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε ανασχηματισμό και αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και με πολύ μεγάλη προσοχή εξετάζουμε και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση στο θέμα αυτό. Αλλά θέλω να σας καθησυχάσω και σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι σε όλα αυτά τα θέματα, όπως άλλωστε και στην περίπτωση των χημικών αποβλήτων, όπου ανταποκριθήκαμε στην, ε, στο λαϊκό αίτημα θα κοιτάξουμε με βάση τις ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές για το περιβάλλον και βέβαια θα στηριχθούμε και στη συνεργασία των ε, ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια και σε εσά για να βρούμε μια στέρεη απόφαση. Για τη διαδικασία του Βερολίνου τώρα. Όταν ξεκίνησε το 2014 είχε θεωρηθεί μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Κυρίως γιατί ακολουθούσε μια κίνηση αποσυμπίεση σχέση με την ε, διεύρυνση και νομίζω ότι αυτό βοήθησε και τις σχέσεις Αλβανίας-Σερβίας και πολιτικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από ότι πριν ε, από τέσσερα χρόνια. Ήδη έχουμε τις δύο πρώτες περιφερειακές πρωτοβουλίες, ε, το, γραφείο, το Περιφερειακό Γραφείο Συνεργασίας ε, των Νέων, με έδρα στα Τύρανα και επικεφαλής Σέρβο και αναπληρωτή διευθυντή Κοσοβάρο δείχνει νομίζω πόσο, μεγάλη, πόσο σημαντική μπορεί να είναι η περιφερειακή διάσταση και η παρουσία στην περιφέρεια. Έχουμε ήδη μια αξιολόγηση και έτσι για την περιφέρεια μπορούμε να γνωρίσουμε τι αποτελέσματα θα έχουν μέχρι το 2030 τα μεγάλα έργα υποδομών. Η, εκλογή, η θητεία μας ωστόσο ε, διαρκεί τέσσερα μόνο χρόνια. Ε, θα θέλαμε, όπως πολύ εύλογα έχει πει η καγκελάριος Μέρκελ, να δούμε περισσότερα έργα να υλοποιούνται στη χώρα. Συνδεσιμότητα πάνω απ' όλα και ουσιαστικά αποτελέσματα για τον πολίτη. Η προσεχή σύνοδος στη Βουλγαρία, σύνοδος κορυφής, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ε, περιφέρεια ολόκληρη και για τις μεταρρυθμίσεις και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αφενός Δυτικών Βαλκανίων αφετέρου Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν παράγον ενίσχυσης ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλεια η ζώνη των Δυτικών Βαλκανίων όταν αντιμετωπίσαμε την μεταναστευτική κρίση ή τους, ε, τις απειλές ε, της τρομοκρατίας, ε, του βίαιου εξτρεμισμού τώρα έχει έρθει η ώρα για μια ε, πιστική λύση στα προβλήματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ε, η χρονική στιγμή θα έχει τεράστια σημασία και βεβαίως πιστεύουμε ότι για τη χώρα μου αλλά και τη Μακεδονία που αναζητά και εκείνη ένα χρονοδιάγραμμα ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκκίνηση των συνομιλιών. Επίσης για την προσεχή σύνοδο και στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, του Λονδίνου, που θα γίνει στο Λονδίνο, η εστίαση θα γίνει θα δοθεί στην ασφάλεια και βέβαια τον ενδιαφέρον που έχει δείξει και το Λονδίνο για το δικό μας το δρόμο, το βαλκανικό δρόμο. Δεν συνεργαζόμαστε την ιδέα αυτή, αλλά ταυτόχρονα και από την άλλη θα προτιμούσαμε να εμβαθύνουμε το τομεί συνεργασίας που έχουν ήδη ξεκινήσει με τη διαδικασία του Βερολίνου, ενέργεια δηλαδή, περιφερειακό οικονομικό χώρο, μεταφορές. Τρεις τομείς που θα έχουν και αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έχουμε ακόμα μερικά λεπτά. Ο Φλέκενστάιν. Knut, du Oh, I will, I will surprise you, so I speak in English. Uh. Θα σας εκπλήξω, θα μιλήσω αγγλικά. Τώρα αγγλικά, μετά ρουμάνικα. Ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Σόλτες. Δεν σας κρύβω ότι πραγματικά με απογοήτευση είδαμε όταν μετά από τόσες συζητήσει ε, στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό και ούτε καν λάβαμε απάντηση. Φυσικά η δική σας κυβέρνηση θα αποφασίσει τι θα κάνει. Θα αποφασίσει λοιπόν τι θα κάνει για αυτό το Εθνικό Πάρκο Ιδρυμό. Όμως σας ε, παροτρύνω να το σκεφτείτε, γιατί αυτή η απόφαση δεν πρόκειται να αναστείλει την πρόοδο, μπορεί να φέρει και οικονομική πρόοδο για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα σας. Αυτό είναι μια σύντομη υπενθύμηση. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει, το σημείωσε ο Υπουργός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπουργέ Μπουσάτη, σας ευχαριστούμε. Όπως ανέφερε και ο συγητής, το 2018 θα είναι χρονιά αποφασιστική σημασία ε, για την Αλβανία και εσείς το δείξατε. Προσωπικά μπορώ να ευχηθώ σε εσά και την κυβέρνησή σας. Καλή τύχη ε, στην προσπάθειά σας να πείσετε τα κράτη-μέλη ότι έχει έρθει η ώρα να ανοίξουν τα πρώτα κεφάλαια, να ξεκινήσουν επισήμως οι δραματεύσεις. Ξέρετε ότι εμείς ειδικά σε αυτή την Επιτροπή είμαστε υπέρ της διεύρυνσης, αλλά βέβαια αυτό εναπόκειται στα 28 κράτη-μέλη. Πρέπει να το αποφασίσουν ομοφόνος. Υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις βέβαια, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και στήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα Δυτικά Βαλκάνια για την Ήπειρό μας και αν δεν εξαγάγουμε σταθερότητα προς τα Δυτικά Βαλκάνια, τότε η πιθανή αστάθεια στα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να ε, ε, ζημιώσει και την Ευρώπη. Γι' αυτό και στηρίζουμε αυτές τις έξι χώρες. Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε στα τύρινα θα θέλαμε να δούμε πόσο καλά συνεργάζεται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Κάποιες φορές ακούω ακόμα ότι υπάρχουν ε, διχογνωμίες και εύχομαι καλή επιτυχία στην κυβέρνηση σε ό,τι φορά την καταπολέμηση των ε, εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε στα διάφορα. Δεν βλέπω κάτι. Επόμενη συνεδρίαση 11 Δεκεμβρίου στις ε, 7.30 έως 9, πέρα συνεδρίασης. We will start the enlarged bureau meeting in 10 minutes. Το διαβριμένο προεδρείο ξεκινάει σε 10 λεπτά στις 6.30.